Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε όλες και όλοι. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν εγκρίνοντας την ημερήσια διάταξη. Έχετε κάποια σχόλια, έχετε παρατηρήσεις, αντιθέσεις όσον αφορά την ημερήσια διάταξη, όχι. Πολύ ωραία, επομένως η ημερήσια διάταξη έχει εγκριθεί. Έχετε λάβει επίσης τα πρακτικά των συνεδριάσεων των 12 και 13 Απριλίου 2011, 2 Μαΐου 2011 και 24 και 25 Μαΐου 2011. Εάν έχετε παρατηρήσει όσον αφορά αυτά τα πρακτικά, παρακαλώ να τις υποβάλλετε στη γραμματεία πριν το πέρας της συνεδριάσεώς μας. Σε αντίθετη περίπτωση θα εγκριθούν τα πρακτικά. Όσον αφορά το σημείο 3, ε, για την ώρα των ερωτήσεων δεν έχουμε κάποια ερωτήματα, επομένως περνάμε και το σημείο αυτό. Όσον αφορά το σημείο 4, ανακοινώσει Προέδρου, δεν έχω να ανακοινώσω οτιδήποτε και επομένως φτάνουμε αμέσως στο επόμενο σημείο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να κάνει κάποιες ανακοινώσεις. Όχι, λέει ο εκπρόσωπος της Επιτροπής. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αλλά παρόλα αυτά δεν έχουμε καμία ανακοίνωση. Eh bien, donc, nous allons passer au vote. Θα περάσουμε στις ψυχοφορίες, λοιπόν. Pardon Oui, mais l'heure, c'est Ça commence à 3 heures. Κοιτάξτε, γιατί να περιμένουμε. Είναι 3 και 5 ήδη. Η ώρα είναι ώρα. Δεν έχουμε εδώ ακαδημαϊκά τέταρτα. Και εάν δεν ξεκινήσουμε αμέσω, λέει η πρόεδρο, κραδένοντα το σφυρί τη, δεν θα τελειώσουμε και στην ώρα μα. Και δεν δίνουμε και το καλό παράδειγμα. Hein? Mais oui, mais bon. On va pas se tourner les pouces pendant 10 minutes non plus. Ναι, και τι θα κάνουμε, θα σταματήσουμε 10 λεπτά. Λοιπόν, έχετε μαζί σας ε, τις κάρτες της ψηφοφορίας σας σε περίπτωση που χρειαστεί ε, να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Να δούμε κάνει. Euh, λοιπόν, για να γεμίσουμε λίγο το χρόνο, επειδή δεν τραγουδάω ωραία, <laughs> λέει η Πρόεδρος, σας προτείνω να ε, ελέγξουμε, να κάνουμε μια δοκιμή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Παρακαλώ ψηφίστε, να δούμε αν λειτουργούν όλα καλά. Άρχεται η ψηφοφορία. Γιατί είχαμε ένα προβληματάκι τεχνικό προλίγου. Μετράω λοιπόν ποιοι έχουν ψηφίσει. Λείπει μία ψήφο. Δεν λέει η Πρόεδρος από πού. Κάποιο συνάδελφο δεν έχει ψηφίσει. Ωραία, λειτουργεί. Ακόμα δεν είναι τρεις και τέταρτο. Τρία λεπτάκια χρειάζονται ακόμα. Ναι, ναι, να μας τραγουδήσετε λοιπόν. Α, εδώ όμως έχουμε και μια τραγουδίστρια. ναι. Κυρία Γκέρεν, θέλετε, θέλετε να μας κάνετε μια ελεύθερη ανάπτυξη θέματος για τρία λεπτά. Euh, Κοιτάξτε, εγώ έχω υποβάλει συγκεκριμένο ερώτημα τραγουδήσετε και εμείς θα χειροκροτούμε μανιωδώς. Donc vous comprendrez que je suis très euh, sensible. Λοιπόν, όχι δεν θέλω να σας κάνω κακό, γι' αυτό δεν πρόκειται να ανοίξω το στόμα μου. Προτιμώ να μην σας κάνω κακό. Την άλλη φορά να βάλουμε τις ψηφορίες λίγο πιο αργά γιατί είναι ανόητο να χάνουμε έτσι χρόνο τουλάχιστον έχει χρόνο να καταφτάσει και ο κύριος Κάσμαν. Τρία λεπτά κύριε Κάσμαν πρέπει να γεμίσουμε το χρόνο. Τα εξής δύο. Μόνο σας περιμέναμε βασικά. <laughs> En tout Encore une minute. Ένα λεπτό ακόμα. du coup, tout le monde arrive. Alors, ceux qui viennent d'arriver, n'oubliez pas de sortir vos cartes de vote. Λοιπόν, για αυτούς που έφτασαν τελευταίοι, παρακαλώ πολύ να έχετε έτοιμες τις κάρτες σας και αν τις έχετε λησμονήσει, θα πρέπει να πάτε να τις ψάξετε, να τις βρείτε, να τις φέρετε. Bon, ben là, c'est bon, hein. Il est 15h15, nous allons voter dans... Λοιπόν, είναι 15 και 15, η ψηφοφορία αρχίζει ακριβώς σε ένα λεπτό από τώρα. Alors, nous allons voter sur euh, le... Θα ξεκινήσουμε λοιπόν την ψηφοφορία στο σχέδιο γνωμοδότησης, για το σχέδιο γνωμοδότησης. Ah, ben, euh, Καταπολέμηση της παράνομης αλληλείας σε παγκόσμιο επίπεδο ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ψηφίσουμε λοιπόν άμεσα από τη στιγμή που δεν είναι το σχέδιο γνωμοδότησης, από τη στιγμή <clears throat> που δεν υπάρχουν τροπολογίες με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Non, mais électronique, pardon. Ηλεκτρονική ψηφοφορία, λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. 20 υπέρ, 20 κατά. Επομένως γίνεται... 20 υπέρ, συγγνώμη συγχαίρουμε τον εισηγητή. Δεύτερο σχέδιο γνωμοδότησης αναβάθμιση της ευρωπαϊκής αντιμετώπισης καταστροφών, ο ρόλος της πολιτικής προστασίας και η ανθρωπιστική βοήθεια. Και εδώ θα έχουμε ονομαστική... Α, θα, ναι, ναι, τελικά θα ψηφίσουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία, αλλά πρώτα τις τροπολογίες. Τροπολογία 1, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρας της ψηφοφορίας. je attendre Non mais c'est bon, on va la rajouter. Hein. Εντάξει, θα μετρήσουμε και τη δικιά σας ψήφο. Εγκρίθηκε η τροπολογία 1, τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές,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 Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στην ηθηγήτρια.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 Amendement numéro 1. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 1, ε, 1, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2, καταπίπτει. Τροπολογία 4, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές. Δεν μέτρησα καλά. Επαναλαμβάνουμε. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 7 <clears throat> υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ κατά Νομίζω ότι θα κάνουμε ηλεκτρονική απαλήθευση. Τροπολογία 10 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 12, όχι, πάμε απευθείας στη 13, τροπολογία 13 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται, τροπολογία 14 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 2, Έχουμε την προφορική τροπολογία υπαριθμών 3 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 15 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβασμός 7 που καλύπτει τις τροπολογίες 16 και 17 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 18 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβασμός 3, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 19 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Α, συγγνώμη, το 19 είχε καταπέσει. Α, μάλιστα. Έπρεπε να μου το πείτε πιο πριν. Τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 25 υπέρ κατά δεν είμαι βέβαια για το αποτέλεσμα. Θα πρέπει να υπαλληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία 25. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ε, ψήφισε ένα ΕΛΚ παραπάνω. Πρέπει να ξαναρχίσουμε. Έχουμε μία ψήφο ΕΛΚ παραπανίσια. Ένα δεν πρέπει να ψηφίσει. από το ΕΛΚ. Άρχεται η ψηφοφορία. Τροπολογία 25. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 26 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η επόμενη καταπίπτει. Τροπολογία 26. Όχι, όχι και αυτή καταπίπτει. Για φαντάσου. Λοιπόν, τροπολογία 30 επομένως λέει η Πρόεδρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ε, νομίζω ότι έχετε μια διαφορά φάσης όταν ψηφίζετε, λέει η Πρόεδρος. Ε, υπέρ. Υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Compromis 4 qui est pour. <laughs> Ένα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Amendement 32. Τροπολογία 32. Τροπολογία 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 5. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 33 καταπίπτει. Η τροπολογία 33 λέει η Πρόεδρος. Όχι, είναι 34. Ε, Πρέπει να μου το λέτε γιατί δεν θυμάμαι τι έχει εγκριθεί και τι όχι. 34, εν πάση περιπτώσει, υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται τροπολογία 35 υπέρ κατά αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβασμός 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 38 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 39 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 40 ε, κατά δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά. Αποχές θα επαληθεύσουμε Δεύτερο τμήμα λοιπόν, η ηλεκτρονική ψηφοφορία, πέρας της ψηφοφορίας, εγκρίνεται. Τροπολογία 41 της παραγράφου 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 42 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 43 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 44 Θέλετε ηλεκτρονική επαλήθευση. Μάλιστα. Προπολογία 43. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ναι, αλλά πρέπει να σηκώνετε τα χέρια σας, λέει η πρόεδρος. Και εγώ κουρασμένη είμαι σήμερα, αλλά τα σηκώνω. 44. Υπέρ. Κατά αποχές Κύριε Κάσμαν, με ένα χέρι θα ψηφίζετε. Ένα χέρι θα σηκώνετε, όχι δύο. Πάντως συγκρίνεται η 44. Παράγραφος 6, τροπολογία 45 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 46 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 2, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 47 καταπίπτει. Άρα τώρα έχουμε την τελική ψηφοφορία. Τελική ψηφοφορία λοιπόν με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίθηκε ομόφωνα συγχαρητήρια στη συντάκτρια της γνωμοδότησης. Άρα. Ε, le Έρχεται η κυρία Γεωργίεβα. Μέχρι να φτάσει όμως θα ζητήσω από την κυρία Βάλστρομ και τον κύριο Όξλεϊ, να, μια και έχουν φτάσει ήδη, να έρθουν κοντά μου. Ah, uh, uh, Merci de reprendre votre place. Ωραία, ξανακαθόμαστε λοιπόν όλοι για να συνεχίσουμε αυτή τη συνεδρίαση. Monsieur Tom, Monsieur Tom. S'il vous plaît, un tout petit peu de silence. Φτάνουμε τώρα στο σημείο 9, πρόληψη ή αντιμετώπιση των ε, καταστροφών, η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την μείωση των κινδύνων καταστροφών. Για αυτήν την ανταλλαγή απόψεων με μεγάλη χαρά ε, θα έχουμε μαζί μας την Επίτροπο κυρία Γεωργίεβα και την κυρία Μαργαρέτα Βάλστρομ, ειδική εκπρόσωπο της Γενικής, του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών, καθώς επίσης και του κύριο Όξλη, ο οποίος είναι εκπρόσωπος της υπηρεσίας ε, τη ε, της πολιτικής προστασίας για τη μείωση των καταστροφών. Έχετε ήδη ε, το, την ημερήσια διάταξη από την προηγούμενη εβδομάδα. Τρία είναι τα γενικότερα ερωτήματα. Τα τρία ερωτήματα λοιπόν, τα οποία τίθενται και γύρω από τα οποία θα περιστραφεί η συζήτηση, είναι τα Ηνωμένα Έθνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτουν τα απαραίτητα εργαλεία έτσι ώστε να εφαρμόσουν τους ε, απαραίτητους μηχανισμούς, τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την πρόληψη των καταστροφών. Δεύτερο ζήτημα, η οικονομία των καταστροφών, πώς μπορούμε να ε, ε, ξοδέψουμε περισσότερα και με καλύτερο τρόπο Επίσης, επόμενη ερώτηση, τι μπορούμε να κάνουμε, ποιο ρόλο μπορούν και οφείλουν να παίξουν ε, οι κυβερνήσεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος και να αντιμετωπιστούν καλύτερα οι καταστροφές. Ε, έχω, έχουμε ζητήσει από τους τρεις παρεμβαίνοντας να ασχοληθούν ε, με τα τρία αυτά ερωτήματα από τη δικιά του σκοπιά ο καθένας θα δώσουμε αμέσως το λόγο στον καθένα από τους καλεσμένους μας για τρία λεπτά. Για δέκα λεπτά, συγγνώμη. Κυρία Επίτροπε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Στα αγγλικά, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας για την ευκαιρία που μας δίνετε να έχουμε σήμερα αυτή τη συζήτηση και ιδιαίτερα παρουσία της Μαργαρέτα Βάλστρομ και του Μάρκους Όξλεϊ. Μόλις ε, συζητούσαμε το γεγονός ότι τους τελευταίους μήνες ήταν πολύ μεγάλη η όθηση για να δοθεί ε, περισσότερη σημασία στο θέμα της μείωσης των ε, καταστροφών. Και θα πρέπει να είμαστε ευγνώμονες στη μητέρα φύση, διότι ήταν πάρα πολύ δύσκολος αυτός ο χρόνος, ε, αυτός ο καιρός, παντού. Πέρυσι αφορούσε ε, αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά φέτος δυστυχώς ανεπτυγμένες χώρες. Άρχισε από την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία που πάλι τώρα επλήγει το Σαββατοκύριακο. Στη συνέχεια είχαμε την Ιαπωνία και τις Ηνωμένε Πολιτείες. Και αυτό που βλέπουμε τι είναι. Δεν μπορούμε πλέον να μιλούμε για ε, μείωση του κινδύνου από ε, καταστροφές στο μέλλον. Είναι κάτι που θα πρέπει να μας απασχολεί τώρα. Είναι στην πολιτική ατζέντα, στην ημερήσια διάταξη των πολιτικών. Και όχι σήμερα από χτες, μάλιστα. Κυρία Πρόεδρε, ακολουθώ την καθοδήγησή σας και θα απαντήσω στις ερωτήσεις, αλλά να αρχίσω πρώτα από ε, τα ε, θέματα της οικονομίας και για την πρόληψη των καταστροφών. Γιατί είναι και οικονομικό το ζήτημα της αδυναμίας μας. Μελέτη, τι μελέτη, τι μελέτη, τι βλέπουμε. Ότι οι επενδύσεις στην πρόληψη και στην ετοιμότητα πιάνουν περισσότερο τόπο από οποιαδήποτε άλλη επένδυση και δημόσια και ιδιωτική σε αυτό το τομέα. Η Παγκόσμια Τράπεζα, πρώην εργοδότης μου, ανακοινώνει ότι για κάθε δολάριο, έστω και ευρώ το ίδιο ισχύει, ε, δεν έχει σημασία το νόμισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επενδύουμε εκεί, η απόδοση είναι 4 με 7 ε, ευρώ ή δολάρια. Δηλαδή είναι 400 με 700% η απόδοση. Και εγώ δεν ξέρω πολλές επενδύσεις που να αποδίδουν τόσο πολύ ε, στον κόσμο. Παρ' αυτά, αν παρατηρήσουμε τι συμβαίνει, και πώς αντιμετωπίζουμε την κατάσταση αυτή. Μας εκπλήσει το γεγονός ότι δεν τα πάμε και τόσο καλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να σας μιλήσω για το θεσμικό όργανο που εγώ εκπροσωπώ. Έχουμε 6 με 8 δις ε, ε, ανάλογα με τη μεθοδολογία που ακολουθούμε ε, για τον υπολογισμό στα διαρθωτικά ταμεία που απευθύνονται άμεσα εκεί, στην ετοιμότητα και την πρόληψη των φυσικών καταστροφών. με δομή αντίστοιχη με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, το, ο κύριος Όγκος πηγαίνει στην αντιμετώπιση των πλημμυρών. Αλλά είναι πολύ χαμηλή η απορρόφηση. Ε, χαμηλότερη, εν πάση περιπτώσει, από άλλη απορροφήση των διαφορετικών ταμείων συνολικά. Δηλαδή, μέχρι τώρα έχουμε χρησιμοποιήσει λίγο περισσότερο από 20% των χρημάτων που είναι στη διάθεση των κυβερνήσεων για να προστατεύουν τον πληθυσμό τους από τους κινδύνους θεομηνιών. Και κάτι άλλο που ενδιαφέρει πάρα πολύ τη δική σας Επιτροπή. Όταν μιλούμε για ε, επενδύσεις ε, στον αναπτυξιακό τομέα, και πάλι μπορούμε, αν θέλετε, να διαφωνήσουμε για τη μεθοδολογία, αλλά μόνο μισό της εκατό της αναπτυξιακής βοήθειας ε, αναφέρεται εκεί και αφιερώνεται εκεί. Την περασμένη εβδομάδα μάλιστα ήμασταν με την κυρία Βάλστον στο Όσλο και ένα από τα συμπεράσματα που βγάλαμε ήταν ότι θα πρέπει να αυξηθεί η συνειδητοποίηση εκείνων που ασχολούνται με την ε, αναπτυξιακή βοήθεια για να καταλάβουμε ποιο τρόπο μπορούν να συμπεριλάβουν στις ε, εργασίες τους και αυτό το στοιχείο, αυτή την πτυχή. Και έρχομαι στο επόμενο ερώτημα, κυρία Πρόεδρε. Τι μπορούμε να κάνουμε για να αυξήσουμε τις επενδύσεις μας στη μείωση των κινδύνων ε, από τις ε, θεομηνίες. Θέλω να σας πω τα εξής τρία σημεία. Πρώτον, να καταλάβουμε καλύτερα τους κινδύνους και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να αντιμετωπίζονται. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε κάνει δύο κινήσεις ή δύο βήματα, αν θέλετε, προς την κατεύθυνση αυτή. Πρώτον, καλέσαμε τα κράτη-μέλη να καταγράψουν τους κινδύνους που τα αφορούν, έτσι ώστε μέχρι το τέλος του 12 να έχουμε μία επισκόπηση και συνολική εικόνα των μεγάλων κινδύνων που απειλούν την Ευρωπαϊκή Ένωση από πλευράς θεομηνιών για να έχουμε μια ε, στρατηγική, ρεαλιστική, επενδυτική στρατηγική ενώ για την αντιμετώπιση. Το ίδιο υποστηρίζουμε και στα προγράμματα για τις αναπτυσσόμενες χώρες, μια καταγραφή ε, του κινδύνου. Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετείχε ε, ως πολύ μεγάλος δωρητής σε ένα πρόγραμμα της Παγκόσμιας Τράπεζας, μια ειδική διευκόλυνση για ε, τα θέματα αντιμετώπισης των καταστροφών. 60 εκατομμύρια ευρώ δίνουμε εκεί και βλέπουμε πως η συλλογική δράση ε, του ΟΗΕ, των Διεθνών Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κάποιων κράτων μελών μαζί μπορεί να προωθήσει την κατανόηση των μεγάλων κινδύνων ε, θεομηνιών στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ήδη έχουμε εντοπίσει 31 προφίλ κινδύνου, θέλετε, για τις πιο ευάλωτες αναπτυσσόμενες χώρες και είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, ήδη από εμά για να μπορούμε να διοχετεύουμε εκεί τη χρηματοδότησή μας για την πρόληψη πάντα των κινδύνων. Στις δικές μου υπηρεσίες, δε, επί σειρά ετών, έχουμε ένα μικρό πρόγραμμα που ονομάζεται Deep Echo. Η Παγκόσμια Τράπεζα, ε, τράπεζα ξέρετε ότι συνεργάζεται με κυβερνήσεις. Εμείς με τοπικές κοινότητες, με πιλωτικά προγράμματα για να έχουμε την εμπειρία ε, από τη βάση προς την κορυφή και να σχεδιάζουμε καλύτερα την πολιτική μας. Με στόχους πάντα τις χώρες που είναι πιο ευάλωτες και πιθανόν να πληγούν περισσότερο. Το δεύτερο βήμα είναι οι ολοκληρωμένες επενδύσεις, δηλαδή ε, κοιτούμε τις υποδομές, την παιδεία, τη δημόσια υγεία, όλους τους τομείς που ε, μπορεί να συνδέονται με τη συνειδητοποίηση και τη δυνατότητα αντιμετώπισης θεομηνιών λάρων καταστροφών. Τώρα με την κλιματική αλλαγή και τη συζήτηση που γίνεται γύρω από αυτή βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή. Επιτέλους, επιτέλους στο Μεξικό είδαμε να αναγνωρίζεται το γεγονός ότι αυτό το θέμα για την κλιματική αλλαγή δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ε, από πλευρά συγκράτηση ή περιορισμού. Έχει φύγει αυτό το τρένο, το έχουμε χάσει. Αυτό που συζητάμε πλέον είναι πώς θα ζήσουμε με τη δεδομένη κλιματική αλλαγή και πώς ε, θα εφαρμόζουμε τα συγκεκριμένα εργαλεία. Γιατί ε, το 90% των θεομηνιών συνδέονται με ακραία φυσικά και καιρικά φαινόμενα. Και επίση θα επέμενα πάρα πολύ ότι θα πρέπει να ξανασκεφτούμε την αιρεσιμότητα των επενδύσεων. Δηλαδή, γιατί θα πρέπει να αφιερώνουμε κονδύλια των φορολογουμένων πολιτών μας σε χώρες που δεν έχουν κάνει τα απαραίτητα βήματα για να μειώσουν τον κίνδυνο ε, να πληγούν από κάποια θεομηνία. Αλλά θα πρέπει να τους πούμε ότι αν θέλετε κοινοτικά κονδύλια επενδύστε πρώτα εσείς αν θέλετε δηλαδή κονδύλια για την αποζημίωση από το Ταμείο Λιλεγγύης κλπ, επενδύστε πρώτα στην πρόληψη. Έχει γίνει λοιπόν μεγάλη συζήτηση για αυτό το θέμα της αρισιμότητας, conditionality, ότι δεν είναι καλό, θα πρέπει να είναι σε αναπτυσσόμενες χώρες, αναχώρα κτλ. Μα σε τελική ανάλυση πρόκειται για την ασφάλεια των πολιτών και ε, έχει και αυτό το στοιχείο το ρόλο του. Και το τρίτο είναι πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα σημεία των αγορών. Παράδειγμα, ασφάλεια. Υπάρχουν χώρες που έχουν χρησιμοποιήσει τις ασφάλειες, τις ασφαλιστικές εταιρείες ε, εκ των προτέρων. Ας πούμε, όταν πρόκειται να χτιστεί ένας οικισμός, ε, ρωτούν ε, τις ασφαλιστικές εταιρείες και δίνουν τη γνώμη τους αν για κατά πόσο είναι επικίνδυνο Χρειάζεται λοιπόν καλύτερο σχεδιασμός για να μειώνεται το κόστος και για την κοινωνία. Δεν ε, χρησιμοποιείται αρκετά αυτό το εργαλείο, ε, έχουμε εκεί υπό Και το τρίτο που είπατε, πώς μπορούμε να αυξήσουμε τη συνειδητοποίηση του κοινού και να τονώσουμε την πολιτική βούληση. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμείς δίνουμε έμφαση στις εξή τρεις δράσεις. Πρώτον, ακριβώς συνειδητοποίηση. Τώρα είμαι εδώ ενώπιόν σας, αλλά εκτός αυτού συνεχώς ταξιδεύω και μπορεί να το μαρτυρήσει αυτό και η κυρία Βάλστρομ ότι με βλέπει πολύ συχνά σε συνεδριάσεις, ιδιαίτερα με εκείνους που σχεδιάζουν ε, την αναπτυξιακή βοήθεια για να τους κάνουμε να καταλάβουν γιατί θα πρέπει να είναι αναπόσπαστο στοιχείο του σχεδιασμού και αυτή η πρόληψη και η μείωση των κινδύνων ε, των ομιλιών. Είναι προτεραιότητα για τη συνεργασία μας και με τον Επίτροπο κύριο Πίμπαλξ και θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι και στις δικές του υπηρεσίες είναι εξίσου ισχυρή δέσμευση με τη δική μας. Γιατί εκεί βλέπουμε πραγματικά εκ των υστέρων τι συμβαίνει όταν δεν έχει κανείς επενδύσει στην πρόληψη. Η συνειδητοποίηση λοιπόν θα πρέπει να γίνει ένα εργαλείο πολύ πιο αποτελεσματικό και να αφορά όχι μόνο εκείνους που ασκούν πολιτική και παίρνουν τις αποφάσεις, αλλά και τους απλούς πολίτες, να καταλάβουν ότι ο κόσμος έχει αλλάξει. Και σε αυτό το νέο κόσμο και για τα παιδιά μας και για τη δική μας ευημερία θα πρέπει ε, να επιμένουμε σε αυτό που κάνουμε με πρόσοχη. Ε, στη συνέχεια, αναλάβαμε κάποια πρωτοβουλία για την οριζόντια ή εγκάρσια συνεργασία μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή αυτό που ε, ζητούμε να κάνουν οι άλλες χώρες θα πρέπει να το κάνουμε κι εμείς. Έχουμε διαπιστώσει ότι το χαρτοφυλάκιο 24 παρακαλώ επιτρόπων συνδέεται με τον ΑΒ τρόπο ε, με αυτό το θέμα της πρόληψης των κινδύνων. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε με ποιους έχουμε άμεσες σχέσεις, άμεσο σύνδεσμο. Άλλες φορές είναι πιο σημαντικός αυτός άλλοτε λιγότερο. Και επίσης οφείλουμε στους πολίτες μας πρέπει να σας πω να προωθούμε πολιτικές ε, με λογοδοσία και σε αυτό το τομέα. Ξέρετε ότι θα φέρω στο Κοινοβούλιο ε, τη στρατηγική μας ε, για τη διαχείριση των θεομηνιών και για την ετοιμότητα και την πρόληψη. Και αυτό που θέλουμε να είναι αυτές οι προτάσεις είναι συγκεκριμένες και όχι ευχολόγια για να έχουμε τα ωφέλη και από τα αποτελέσματα για να δούμε πώς λειτουργεί η οικονομία. Ευχαριστώ κυρία Γεωργίευα. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Βάλστρομ για 10 λεπτά επίσης. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και συνεχίζω στα αγγλικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που μου απευθύνεται. Και εγώ θα δραθώ της ευκαιρίας να ξεκινήσω με τα οικονομικά. Θα σας εξηγήσω γιατί. Όλοι εμείς που έχουμε δουλέψει βάσει της απλής λογικής ότι οι καταστροφές μπορούν να προληφθούν ε, έτσι ώστε να ε, περιοριστεί το κόστος και να περιοριστούν και οι επιπτώσεις επιπτώσεις ε, στους τοπικούς πληθυσμούς. Δουλεύουμε στα θέματα αυτά 30 και καμιά φορά και 40 χρόνια. Ε, αναρωτιόμαστε λοιπόν, όπως και η Επίτροπος κυρία Γεωργίευα, γιατί δεν έχουμε καταφέρει να αλλάξουμε λίγο ε, την αντιμετώπιση και γιατί δεν γίνεται ένας καλύτερος σχεδιασμός. Καταρχήν, ε, βεβαίως το πρώτο που μας απασχολεί είναι η ανθρωπιστική διάσταση. Οι ζωές των ανθρώπων πρέπει να σώζονται και σώζονται και σώζονται περισσότερο και καλύτερα. Το παράδειγμα λοιπόν το σημερινό είναι ότι με σωστή δουλειά μπορούμε να σώσουμε περισσότερες ε, ζωές. Ε, βεβαίως ε, θα πρέπει να δούμε πώς μπορεί κανείς να περάσει από την αντίδραση και την πληρωμή στην προηγούμενη φάση, την πρώτερη φάση, δηλαδή την πρόληψη. Σήμερα έχουμε ε, και μία έκθεση ε, της, ε, ε, των Ηνωμένων Εθνών, μπορείτε να την συμβουλευτείτε κιόλας, σύμφωνα με την οποία οι κίνδυνοι αυξάνονται σε ολόκληρο τον κόσμο. Θα πρέπει να μελετήσουμε τις καταστροφές έτσι ώστε να δούμε ποιοι είναι οι κίνδυνοι οι οποίοι συσσωρεύονται. Ποιοι είναι αυτοί μεγάλη και γρήγορη αύξηση ε, των πληθυσμών που ζουν είτε σε δέλτα ποταμών είτε ε, σε ε, παράκτιες και παρόχθιες περιοχές. Έχει αλλάξει ο πληθυσμός που κατοικούσε ε, στην γη μας ε, ε, σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, αλλά έχει αυξηθεί κατά 92% ο πληθυσμός που κατοικεί σε πάρα πολύ επικίνδυνες περιφέρειες του κόσμου και επομένως αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο για φτωχές χώρες αλλά ισχύει και για τις πιο πλούσιες ε, χώρες. Ε, ο κίνδυνος δεν είναι καλά χαρτογραφημένος ε, γιατί όλες οι χώρες δεν συλλέγουν στοιχεία είτε για τις καταστροφές είτε για τους κινδύνους που συσσωρεύονται. Βεβαίως άνθρωποι που κάνουν τη δουλειά που κάνω και εγώ πάντοτε συμβουλεύουν να υπάρχουν τέτοιοι κατάλογοι έτσι ώστε να αποφεύγεται ο συνοστισμός ας πούμε πληθυσμών ε, σε δέλτα ποταμών και σε ιδιαίτερα επικίνδυνες ε, ε, περιοχές να δημιουργούνται κατάλογοι οι οποίοι θα μπορούν να χρησιμοποιούνται προς αποφυγή κινδύνων. Πάντως μπορώ να πω ότι ο κίνδυνος, όπως είπα και στην αρχή, ε, αυξάνεται ε, σε όλες τις χώρες. Αλλά ο κίνδυνος ίσως είναι και μεγαλύτερος και γρηγορότερα αυξανόμενος για τις πιο πλούσιες χώρες, οι οποίες έχουν πολύ πλούτο να χάσουν και μπορεί η κατάπτωσή τους ε, να είναι πάρα πολύ γρήγορη. Ε, οι χώρες οι οποίες είναι όμως περισσότερο εκτεθειμένες είναι οι χώρες όσα ε, νομίζω ότι σαφώς καταδεικνύεται αυτό από όλες τις μελέτες. Τι απορρέει από αυτή ε, τη διαπίστωση ότι οι χώρες μας δεν κατανοούν ακόμα τον κίνδυνο πρέπει να δοθούν και οικονομικά στοιχεία, αλλά υπάρχουν πολλά οικονομικά στοιχεία, πολλές οικονομικές μαρτυρίες που οδηγούν προς αυτό το ε, θέμα ε, και προς, αυτήν την, ε, προς αυτό το συμπέρασμα. Επομένως, ενδεχομένως, λείπει η πολιτική βούληση. Υπάρχει μία χώρα στον κόσμο η οποία έχει νομοθετήσει ε, την ε, ε, προσωπική λογοδοσία για τους κυβερνώντες οι οποίοι δεν αντιμετωπίζουν σωστά ή δεν προλαμβάνουν σωστά τις καταστροφές. Αυτή η χώρα είναι η Ινδονησία, η οποία βεβαίως είναι πολύ εκτεθειμένη θα πρέπει κανείς να μπορεί να φτάσει στους υπεύθυνου ε, ε, και νομίζω ότι αυτό θα γυρίσει μια νέα σελίδα στην κατάσταση. Ε, δεν δίνονται λοιπόν, δεν δίνεται λοιπόν σωστή ορατότητα στα οικονομικά συστήματα στο κεφάλαιο 5 αυτής της έκθεσης ε, που αναφέρει πολλά μακροοικονομικά στοιχεία που σχετίζονται με τους κινδύνους καταστροφής. Δείχνει στο βάθος της αίθουσας, όπως σας είπα προηγουμένως, είναι το κεφάλαιο 5, μπορείτε να το μελετήσετε μπορούν να υπάρξουν επενδύσεις, μπορούν ε, να χρησιμοποιηθούν πάρα πολλές δυνατότητες είτε επανεπένδυσης χρημάτων, είτε διαχείρισης κινδύνου κτλ. Αυτό μπορεί να γίνει στις ε, ε, φτωχότερες χώρες του κόσμου. Ο Πολύ λιγότερο. Η απάντηση είναι προφανώς αρνητική γιατί ούτως ή άλλως οι πολίτες είναι αυτοί που πληρώνουν τις το περισσότερο ποσό ε, των καταστροφών. Ε, τα Ηνωμένα Έθνη, οι τράπεζες, ε, πολλαπλή φορείς προσπαθούν να διδάξουν στις χώρες πώς να χρησιμοποιούν τα εργαλεία. Και βεβαίως νομίζω ότι εγώ αυτό που μπορώ να πω στους πολιτικούς είναι να χρησιμοποιούν τα στοιχεία και να χρησιμοποιούν την πραγματογνωμοσύνη πραγματογνωμοσύνη τους ε, και εκεί να βασίζονται έτσι ώστε να δημιουργήσουν ε, ένα καλό υπόβαθρο αν μπορούμε να συνεργαστούμε καλύτερα, βεβαίως μπορούμε. Ε, ήδη συνεργαζόμαστε και την Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή. Εμείς ε, πάντα λέμε, προσπαθούμε να βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα στους διεθνεί φορείς, στους εθνικούς φορείς, τους διάφορου οργανισμούς, έτσι ώστε να υπάρχει μια ένα γενικότερο υπόβαθρο. Υπάρχει ήδη από το 2005 ε, μια συνολική αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών επί, των, ε, έχουμε συμφωνήσει ε, πολλοί φορείς. Ένα από τα κυριότερα προβλήματα ε, είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορεί κανείς να ξεπεράσει τα θεσμικά προσκόμματα έτσι ώστε να φτάσει σε ένα επίπεδο το οποίο είναι απαραίτητο έτσι ώστε ε, να ε, αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι δηλαδή πότε οι κυβερνήσεις απευθύνονται στα Ηνωμένα Έθνη, ποιος θα ηγείται κάποιας προσπάθεια, ε, νομίζω ότι θα πρέπει ε, να ε, κρατηθεί αυτή η πολιτική ηγεσία και η ιδέα αυτή, αλλά βεβαίως να υπάρχει και ένα ολόκληρο υπόβαθρο ή ένα δίκτυο το οποίο θα αφορά συνεργασία οργανισμών. Θα πρέπει να γίνεται μια προσπάθεια επίσης να λαμβάνεται υπόψη η πρόοδος που έχει γίνει από άλλους φορείς και είναι γεγονός ότι δεν προοδεύουν όλοι με τον ίδιο ρυθμό. Ε, αυτό που έχω να πω είναι ότι ο κόσμος γενικότερα βλέπει λίγο θαμπά το θέμα της πρόληψης γιατί δεν είναι σαφές. Είναι λίγο ασαφές το τι σημαίνει πρόληψη λέμε ας πούμε ε, στα, παιδιά ότι όταν πλένεις τα χέρια σου τακτικά αυτό θα σε κρατήσει υγιή και για την υπόλοιπη ζωή σου. Ας δούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Ε, διαχείριση των υδάτινων πόρων. Να μάθουμε τον κόσμο να μην ξεχνάει τις φυσικές καταστροφές. Να μαθαίνουμε από τα λάθη μας, να διδασκόμαστε από τα λάθη μας. και όταν έγινε το ατύχημα, μάλλον πριν γίνει το ατύχημα την, της Φουκουσίμα, ε, μου έλεγε ένας ηθήνων της χώρας ότι ε, φοβότανε γιατί ο κόσμος φαινόταν να έχει ξεχάσει τον προηγούμενο μεγάλο σεισμό. Ε, νομίζω λοιπόν ότι ο καθένας στη χώρα του θα πρέπει να διασφαλίζει ότι όλοι οι τεχνικοί φορείς και τομείς ε, αισθάνονται ότι πρέπει να βρίσκονται πάντα σε επαγρύπνηση. Θα πρέπει λοιπόν να έχει η χώρα μια καλή διοικητική δομή, να υπάρχει καλή συνεργασία ε, μεταξύ των διαφόρων φορέων, αλλά βεβαίως να υπάρχει και απαραίτητη χρηματοδότηση. Και φυσικά τα διάφορα τεχνικά σκέλη ε, ε, μιας κυβέρνησης, μιας χώρας να είναι σε θέση να έχουν την απαραίτητη προετοιμασία και τους απαραίτητους μηχανισμούς έτσι ώστε να μπορούν να συντονίσουν καλά την δράση τους ε, θα πρέπει να υπάρχει μια εθνική πλατφόρμα ε, η οποία θα ε, φέρνει γύρω από ένα τραπέζι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που ενδεχομένως δεν μπορούν να παίρνουν αποφάσεις αλλά πάντως θα μπορούν να φέρουν την γνώση, την καλή θέληση και την εμπειρία μαζί. <coughs> Συνεργασία λοιπόν μεταξύ περιφερειακών και εθνικών αρχών, μεταξύ εθνικών αργών, αρχών και διεθνών οργανισμών ε, και ξέρετε ότι ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών ας πούμε έχει πάρει πάρα πολύ σοβαρά ε, αυτά τα θέματα. Τεχνική ικανότητα, καλή ε, θέληση λοιπόν και χρήματα αυτά είπαμε μαζί με την καλή ηγεσία Κοιτάξτε, ε, νομίζω ότι είναι πλέον σαφές ότι οι πολίτες ζητούν περισσότερη ασφάλεια. Όταν οι κυβερνήσεις και οι τοπικές κυβερνήσεις ε, κατανοούν πόσο τρομακτικά κοστίζουν οι φυσικές καταστροφές, ε, τότε πραγματικά θα καταλάβουν γιατί μιλάμε. Γενικώ είναι πολύ εκτεθειμένοι η υποδομή σε ολόκληρο τον κόσμο. Έχουμε ολο ένα αυξανόμενα κόστη λόγω της πίεσης που προκαλεί η αύξηση του πληθυσμού ε, και λόγω της μεγάλης έκθεσης των, ε, των διαφόρων υποδομών ε, σε πολλούς κινδύνους και νομίζω ότι διάφορες φυσικές καταστροφές των δύο τελευταίων ετών μας ε, δίνει ακριβώς να κατανοήσουμε τη μεγάλη διάσταση. Κοιτάξτε, εμείς ζητούμε στην ουσία πολιτικούς ηγέτες, πολιτικούς οι οποίοι να μπορούν να παίξουν ηγετικό ρόλο ε, και σε τοπικό επίπεδο όπως ας πούμε ο δήμαρχος της πόλης του Μεξικό με μονομένοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο ε, έτσι ώστε να γίνει κατανοητή η σημασία της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων. Έχουμε επίσης τα παιδιά τα οποία ζητούν και απαιτούν καλύτερη δράση και καλύτερη αντιμετώπιση. Ε, εμείς καταφέραμε επίσης να κινητοποιήσουμε τον πρόεδρο της ε, Ινδονησίας έτσι ώστε στην δικιά του περιοχή να προωθήσει αυτή την ατζέντα. Γιατί το μήνυμα είναι πάρα πολύ σαφές, όσο και απλό. Όταν θα πάμε στο Ρίο του Τζανέιρο του χρόνου, να συναντηθούμε, να δούμε τι καταφέραμε όσον αφορά ε, την βιώσιμη ανάπτυξη τα τελευταία 20 χρόνια. Εάν δεν λάβουμε υπόψη μας τους δύο-τρεις σημαντικούς κινδύνους στη βιώσιμη ανάπτυξη, δηλαδή φυσικές ε, καταστροφές, κλιματική αλλαγή και ανικανότητά μας να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της φτώχειας παγκοσμίως, τότε δεν θα έχουμε καταφέρει και πολλά όσον αφορά ε, την ε, βιώσιμη ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα τον λόγο στον κύριο Μάρκους Όξλεϊ. Για 10 λεπτά παρακαλώ. 10 um, uh, Δέκα λεπτά μου δώσατε για τις ερωτήσεις που είναι στο έγγραφο και θα σας πω λίγα πράγματα από τη σκοπιά της ε, μιας οργάνωσης δηλαδή της κοινωνίας των πολιτών με 600 οργανώσεις υπό την αιγίδα μας που εργάζονται στο τοπικό επίπεδο από 90 χώρες και θα σας ε, αναπτύξω λοιπόν τις, ε, τις θέσεις αυτές. Όταν μιλούμε για DRR, κατά τη γνώμη μου, αυτό δηλαδή που καταλαβαίνω, είναι ένας τρόπος για να κάνουμε αναπτυξιακή δουλειά σε ένα χώρο, σε ένα τομέα όπου ε, υπάρχουν κίνδυνοι, είτε πρόκειται για δημόσια επένδυση είτε για άλλα πράγματα. Δηλαδή για το πώς επενδύουμε στον τομέα αυτό ή στο έργο αυτό σε μια περιοχή η οποία έχει κινδύνους. Στα πλαίσια ενός κλίματος που αλλάζει όλο και περισσότερο. Αυτή λοιπόν είναι η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε. Πώς κάνουμε αναπτυξιακή δουλειά σε ένα χώρο κινδύνου και εάν μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα αυτό θα έχουμε απόδοση των επενδύσεων. Δηλαδή την απόδοση των επενδύσεων που επιθυμούμε να έχουμε. Στο τοπικό επίπεδο από την σκοπιά των τοπικών οικοκυριών ο κόσμος δεν κάνει διάκριση ανάμεσα στους θεματικούς αυτούς τομείς, δηλαδή προσαρμογή στο, στην αλλαγή του κλίματος, ε, στην κρίση, όλα από τη σκοπιά τους είναι ένα συνολικό πρόβλημα. Προστασία των ανθρώπων, ασφάλεια, προστασία της ε, ευημερία τους, ευημερίας τους, του επίπεδου, των ε, στοιχείων ενεργητικού τους, της περιουσίας τους εν τέλει. Ε, εγώ είμαι μηχανικός και βρίσκω ότι form follows function και αυτό που εννοούμε με άλλα λόγια είναι ότι η διάρθρωση των πραγμάτων θα πρέπει να ακολουθεί πρωτίστως τον σκοπό που ε, η δομή αυτή επιδιώκει να επιτύχει. Δηλαδή για το πρώτα, για να, για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις δομές, πρώτα θα πρέπει να έχουμε υπόψη τι θέλουμε να επιτύχουμε στο τοπικό επίπεδο. Και το πρόβλημα είναι, τα προβλήματα μάλλον είναι αλληλοσυνδεόμενα και δεν χωρίζονται σε αυτούς τους θεσμικούς πυλώνες που μετά το πρόβλημα είναι πώς θα τους εντάξουμε σε ένα όλον. Ενώ στην ουσία έχουμε αυτή την νοοτροπία ότι όλα είναι ξεχωριστά. Γιατί στο τοπικό επίπεδο τα πράγματα είναι παρόμοια. Δηλαδή, αν επιθυμούμε να βελτιώσουμε τις δομές μας και τους θεσμικούς μηχανισμούς μας, νομίζω θα μας βοηθήσει αν έχουμε ένα συνολικό πλαίσιο σχεδιασμού που περιλαμβάνει και αυτά που λέμε resilience, ανθεκτικότητα δηλαδή, και σε ακραίους κινδύνους, αλλά και στις πιο σταδιακές αλλαγές για παράδειγμα τις κλιματικές αλλαγές που αρχίζουμε και βλέπουμε και που έχουν πιο αργούς ρυθμούς. Όταν εξετάσουμε λοιπόν πώς ε, θεμελιώνουμε αυτή την ανθεκτικότητα στο τοπικό επίπεδο θα δούμε ότι τα πράγματα είναι πολύ παρόμοια. Είτε δηλαδή μιλούμε για θέματα αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών, είτε της μείωσης των κινδύνων, είτε την ελάφρυνση της φτώχειας. Διαπιστώνουμε ότι τα βασικά συστατικά που ε, η προσπάθειά μας είναι να δώσουμε στο τοπικό επίπεδο είναι να μπουν οι άνθρωποι στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, να βασιστούμε στις τοπικές ικανότητες, τεχνογνωσία, δηλαδή να βασιστούμε στις ικανότητες των ίδιων των ανθρώπων, οι άνθρωποι να έχουν πολιτική κυριότητα εντός εισαγωγικών των ε, ε, όσων συμβαίνουν επί τόπου, όχι δηλαδή να έρθουμε εκ των άνω να τους επιβάλλουμε την ε, ανθεκτικότητα αυτή. Πρέπει να υπάρχει μια, ένα αίσθημα ότι αυτοί είναι οι ιδιοκτήτες της υπόθεσης. Και μία από τις αρχές που χρησιμοποιούμε για να φτιάξουμε αυτή την ανθεκτικότητα είναι και, για παράδειγμα, το δικαίωμα της συμμετοχής, το δικαίωμα στην ενημέρωση, το δικαίωμα στην μη διάκριση, το δικαίωμα σε αποζημίωση. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει και μια accountability, μια λογοδοσία σαν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Εσείς βέβαια γνωρίζετε καλύτερα τις θεσμικές σας δομές και διαδικασίες, από ότι, πολύ καλύτερα από ότι τα γνωρίζω εγώ, αλλά αν θέλουμε να τα βελτιώσουμε, ας έχουμε πρώτα υπόψη ποιες ακριβώς αλλαγές θέλουμε να επιφέρουμε στο τοπικό επίπεδο, και ας ε, αντιληφθούμε ότι πολλές ομοιότητες και επικαλύψεις υπάρχουν πραγματικά που νομίζω στο επίπεδο των επιχειρήσεων θα το λέγαμε consolidation και rationalization όπως για παράδειγμα στις συγχωνεύσεις μεταξύ επιχειρήσεων, έτσι θα το λέγαμε, ε, ε, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν σημαντικές επικαλύψεις. Όταν, όταν λοιπόν λέμε τώρα πώς θα αποδώσουν καλύτερα οι επενδύσεις μας, νομίζω ότι αυτά τα πράγματα συνδέονται πολύ στενά. Γιατί μιλούμε για την οικονομική πτυχή των ε, θεομηνιών και καταστροφών ως φορολογούμενοι εμείς εδώ. Πώς θα επιτύχουμε τη μέγιστη απόδοση των επενδύσεών μας, γιατί περί αυτού πρόκειται εν τέλει, έτσι δεν είναι. Δηλαδή πώς θα επιτύχουμε η επένδυσή μας αυτή να έχει στο μάκρο οικονομικό επίπεδο το υψηλότερο δυνατό, την υψηλότερη δυνατή απόδοση. Διαπιστώνω λοιπόν ω κοινωνία πλέον ότι κάνουμε, ω civil society δηλαδή, ότι κάνουμε μια προσπάθεια, βάζουμε τους σχεδιαστέ, του νομοθέτες να συνεργαστούν και όταν οι κυβερνήσει έρχονται και λένε που επιτύχανε κάποια πρόοδο, είναι σαφές, υπάρχουν σαφή στοιχεία στο, στο εθνικό επίπεδο ότι οι πολιτικέ DRR αρχίζουν και ε, μπαίνουν στη θέση τους. Το πρόβλημα είναι αυτό. Τι η νομοθεσία, οι νομοθετικές διατάξεις δηλαδή να μπουν στην πράξη στο επίπεδο, στο τοπικό επίπεδο. Η εκτέλεση δηλαδή της πολιτικής αυτής. Και εδώ από τη δική μου σκοπιά βρίσκεται το κενό μέσα στο σύστημα. Δηλαδή ότι αυτές οι μακροοικονομικές εισρωές δεν έρχονται να φτάσουν στο μικρό επίπεδο. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την απόδοση των επενδύσεών μας, ακόμα έχουμε μεγάλο δρόμο να διανύσουμε για να επιτύχουμε αυτά που θέλουμε. Και νομίζω ότι εδώ επανερχόμαστε σε ορισμένες βασικές αρχές. Δηλαδή τα μετρήσιμα είναι και διαχειρίσιμα. Εάν δηλαδή έχουμε ξεκάθαρα μέσα στο μυαλό μας τι επιθυμούμε να επιτύχουμε στο τοπικό επίπεδο, έχουμε και ξεκάθαρα πλαίσια παρακολούθησης, monitoring επιτόπου, έχουμε δηλαδή διαφάνεια και λογοδοσία στο επίπεδο επιτόπου ότι δηλαδή αυτά που βάζουμε πάνω βγαίνουν κάτω στο, στο χαμηλό, στο τοπικό επίπεδο ότι υπάρχει διαφάνεια δηλαδή για το πού πηγαίνουν αυτές οι χρηματοδοτικές ροές και σε τι μεταφράζονται τελικά νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε ευφιέστερα τους πόρους μας. Και νομίζω ότι οι βασικοί δείκτες είναι όντως στο τοπικό επίπεδο. Δηλαδή, εφόσον οι πολιτικές αυτές δεν επιφέρουν συστημικές αλλαγές στο τοπικό επίπεδο, στις τοπικές αρχές, τοπικές κοινότητες, τοπικές ομάδες, τότε θα μείνουν στα λόγια. Και αυτό που φοβούμε είναι ότι φτιάχνουμε, έτσι λέμε, πολλά ε, στο επίπεδο της πολιτικής ρητορική, αλλά δεν φτάνουμε να αποδώσουμε στο μικρό επίπεδο. Και έρχομαι στο τρίτο σημείο που θέλω να θίξω, η πολιτική δηλαδή βούληση, δηλαδή πώς μεταφέρει κανείς τα λόγια σε πράξεις. Ε, έχω σημειώσει μερικές ιδέες εδώ σχετικά με το πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό, δηλαδή κοινά πλαίσια στο τοπικό επίπεδο που να εναρμονίζουν και να ενώνουν τους θεματικούς αυτούς τομείς για τους οποίους μιλήσαμε να μπουν οι άνθρωποι μέσα στις διαδικασίες, να νιώσουν ότι είναι κύριοι της διαδικασίας, ότι αυτή έχει μια διάρκεια, ότι οι αρχές λοιπόν της συμπερίληψης, της συμμετοχής είναι απόλυτα σημαντικές, ζωτικής σημασίας, θέματα διαφάνειας και λογοδοσίας επίσης είναι κρίσιμη σημασίας επίσης η χρήση των πόρων για να δημιουργηθεί local capacity, για να δημιουργηθούν ικανότητες επιτόπου. Αν δεν έχουμε ικανότητες επιτόπου στο τοπικό επίπεδο, δεν μπορούν τότε οι πολιτικές, τα ωραία λόγια δηλαδή, εν τέλει να μετατραπούν σε πράξεις επιτόπου. Και επανέρχομαι σε αυτό που είπε και η Μαργρέτε, το ζήτημα αυτό της ε, συνειδητοποίησης του κοινού, της, ε, της ε, κοινωνικής αξίωσης, πρέπει να γνωρίζουν οι άνθρωποι ποια είναι τα θέματα ποιες είναι οι υποχρώσεις των κυβερνήσεων, τα καθήκοντά τους. Να γνωρίζει ο κόσμος δηλαδή, να γνωρίζουν οι άνθρωποι συγκεκριμένα ποιες είναι οι πολιτικές, ποιες είναι οι νομοθεσίες. Δεν θα πιω τσάι αυτή τη στιγμή, σας ευχαριστώ. Όχι, ευχαριστώ πολύ. Ορισμένες λοιπόν βασικές ιδέες οι οποίες έχουν σχέση με αυτή την ε, την προβολή αξιώσεων στο τοπικό επίπεδο. Και αυτό νομίζω ότι χρειάζεται ε, πολύ μεγαλύτερη επένδυση στην πλευρά της ζήτησης. Καλά τα καταφέρνουμε από την πλευρά της προσφοράς, αλλά εδώ χρειάζεται να εξασφαλιστεί σωστή ισορροπία ανάμεσα στο εκ των άνω και στο εκ των κάτω. Εγώ δεν λέω ότι πρέπει όλα να είναι εκ των κάτω, ούτε όμως μπορούν να είναι και όλα η πλευρά της προσφοράς και από πάνω προς τα κάτω. Πρέπει να υπάρχει κάποια μέση οδός. Και νομίζω ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε ώστε οι επενδύσεις μας προσφέρουν και όθηση και έλξη. Δηλαδή και από πάνω οθούν αλλά και από κάτω πρέπει να φτιάξουμε, να δώσουμε την ικανότητα στους ανθρώπους να προβάλλουν αξιώσεις, να υπάρχει και η έλξη προς τα κάτω, προς το χαμηλό επίπεδο, προς το μικρό επίπεδο. Και αυτά και στις δικές σας εκλογικές περιφέρειες και στη δική σας πολιτική στράτευση. Αυτό θέλετε να κάνετε, να μπουν οι άνθρωποι μέσα, να συμμετάσχουν, να έχουν την αίσθηση ότι είναι κύριοι της διαδικασίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στους βουλευτές. Θα ξεκινήσουμε την κυρία Θεοχάρους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όλοι οι ομιλητές ξεκίνησαν με μια φιλοσοφική προσέγγιση του ζητήματος και παράλληλα παρουσίασαν και τα πρακτικά μέτρα που εισηγούνται για την πρόληψη για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Όσον αφορά τη φιλοσοφική προσέγγιση, επιτρέψτε μου και εμένα να πω ότι στην φύση, στην βιολογία υπάρχει η αρχή της ισορροπίας, της ομοιόστασης. Η ανεξέλεκτη ανάπτυξη ενός πληθυσμού οδηγεί την φύση να αντιδράσει κατά τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να περιορίσει δραστικά τον πληθυσμό. Και έχουμε, μπορώ να σας δώσω δέκα παραδείγματα αυτή τη στιγμή τέτοιων φαινομένων από την παγκόσμια ιστορία. Δυστυχώς όσο και αν αυτό είναι πεσημιστικό, το ίδιο ισχύει και για τον, το ανθρώπινο είδος. Έχει φτάσει πια σε ανεξέλεκτους αριθμούς και η φύση ίδια θα αντιδράσει. Αν δεν αντιδράσει η φύση και αν δεν υπάρξει μείωση του ανθρώπινου πληθυσμού, σίγουρα θα εξαφανιστεί το ανθρώπινο είδος. Αυτό ας μου επιτραπεί, θα μπορούσα να μιλώ πολλή ώρα για αυτό το θέμα, αλλά ας μου επιτραπεί μια ανάπτυξη, μια προσέγγιση τέτοια. Όσον αφορά τα πρακτικά ζητήματα, ναι. Οι επιπτώσει μπορούν να προληφθούν, όχι όμω οι ίδιες οι φυσικέ καταστροφέ. Και αυτό φάνηκε και από τον σεισμό στη Χιλή, όπου λόγω τη καλή υποδομή στη χώρα δεν είχαμε ίδια ένταση σεισμό, δεν είχε τα ίδια αποτελέσματα όπω είχε στην ΑΙΤ για παράδειγμα. Η ένταση των επιπτώσεων μπορεί να μειωθεί και αυτό πάλι όπω έχετε πει με τη συσσόρευση πληθυσμού στα δέλτα των ποταμών σε ευαίσθητα σημεία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να ελέγξουμε ε, κατά κάποιο τρόπο. Και με τη δημιουργία της σωστής υποδομής στις διάφορες περιοχές του πλανήτη. Το Ταμείο Αλληλεγγύης είναι ένα σημείο στο οποίο εμείς ως ε, Ευρωπαίοι Βουλευτές θα μπορούσαμε να δράσουμε πραγματικά και να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη του. Η παρέμβαση στο επίπεδο της κοινότητας είναι κάτι το συγκλονιστικό για μένα που έχει αναφέρει η κυρία Επίτροπος γιατί πραγματικά επειδή εγώ γνωρίζω πολύ καλά τι σημαίνει η παγκόσμια διαφθορά σε επίπεδο κυβερνήσεων είναι ξεκάθαρο ότι μόνο η παρέμβαση στο επίπεδο της κοινότητας μπορεί να δώσει τη δυνατότητα άμεσης ανάπτυξης και αντιμετώπισης των καταστροφών και χαίρομαι πάρα πολύ κυρία Επίτροπε γι' αυτό που έχετε πει. Η δύναμη ταχεία αντίδρασης είναι κάτι το οποίο απαραίτητα πρέπει να δημιουργήσουμε στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά να συνεχίσουμε τις προσπάθειες. Γιατί θυμάμαι πριν από 10-15 χρόνια ήταν πάρα πολύ της μόδας να αντιμετωπίζουμε το desertification φυτεύοντας δέντρα παντού. Να αντιμετωπίσουμε... Θυμάμαι από την ε, Γκόμπη, την έρημο Γκόμπη, στην εσωτερική Μογγολία, στη ε, Καλαχάρη κλπ. Τώρα αυτά τα πράγματα έχουν σταματήσει γιατί κουράζουν την, ε, του, τους πολίτες και μέσα σε χρονικό, σύντομο χρονικό διάστημα όταν πάψει πια να είναι της μόδας σταματούν να ασχολούνται και με αυτό. Άρα εκείνο που έχετε πει ότι πρέπει να υπάρχει συνεχής και σωστή ενημέρωση είναι επίσης ένα ε, δραματικό σημείο στο οποίο πρέπει να επιμείνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Merci beaucoup. Nous allons poser trois questions à la Τρεις ερωτήσεις ε, κάθε φορά και μετά θα απαντάτε. Ο κύριος παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ βεβαίως με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τους ε, παρεμβαίνοντες ε, του παρακολούθησα τις εισηγήσεις τους με μεγάλη προσοχή και τις θεώρησα εξαιρετικά επικοδομητικές. Θα ήθελα να σχολιάσω αυτά που είπε η Επίτροπος η κυρία Γεωργίευα, η οποία όπως πάντα με πολύ δόκιμο τρόπο μας είπε πόσο σημαντικό είναι να κάνουμε καλή προληπτική πολιτική. Υπογραμμίσατε δε περισσότερο την ε, τύχη ε, σε αυτές τις περιπτώσεις η επιστροφή των επενδύσεων να είναι ιδιαίτερα σημαντική. Έχω να ρωτήσω λοιπόν το εξής μια και σας άκουσα να μιλάτε για πρόληψη ε, κινδύνων και κυρίως την εφαρμογή ε, και κυρίως μάλλον ε, την έμεση ή άμεση συμμετοχή 23 επιτρόπων με τα θέματα αυτά. Το, ρωτώ λοιπόν, έχετε όρια και αν ναι, ποια είναι τα όρια. Και γίνομαι πιο συγκεκριμένο. Η πιο μεγάλη καταστροφή των έξι τελευταίων μηνών ήταν αυτή τη Φουκουσίμα. Ε, συνδέεται λοιπόν άμεσα με την πυρηνική ενέργεια. Ε, τα, ε, τα τεστ προσωμείωσης ακραίων φαινομένων, τα λεγόμενα τεστ ανοχής, έγιναν βεβαίως εν είδη προλήψεως μελλοντικών πυρηνικών ατυχημάτων. Η διηγενική σας διεύθυνση έχει αναμειχθεί στις διαδικασίες αυτές. Έχετε κάτι να μας πείτε όσον αφορά αυτό το θέμα. Ε, δεν θέλω να θέσω κάποιο άλλο ερώτημα, γιατί θεωρώ ότι ήδη είναι αρκετά περίπλοκο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να πω δύο λόγια. Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης ε, μεταξύ των εταίρων ε, για την ανανέωση του νομοθετικού πλαισίου την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, η συνιστόσα της ε, ε, πρόληψης πραγματικά φάνηκε να είναι κυριαρχούσα. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια για τον χώρο που καταλαμβάνει η πρόληψη και να το σχετίσετε με την πρόληψη των καταστροφών και την άμεση αντιμετώπιση των καταστροφών. Θα ήθελα να απαντήσετε και μετά θα κάνουμε άλλες τρεις ερωτήσεις. Είμαι ευγνώμων στην κυρία Θεοχάρους γιατί ακριβώς ανέφερε το θέμα της ε, ε, απερίμωσης, το θέμα της ε, καταστροφής των δασών. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την χιλή και την τεράστια επένδυση που έκανε η χιλή ως σεισμογενής χώρα έτσι ώστε να σταθεροποιήσει τα πρανή των ε, ε, βουνών και βεβαίως και ε, να προλάβει τον κίνδυνο. Η αποψήλωση δεν είναι μονάχα, δεν αποτελεί απειλή μονάχα για χώρες οι οποίες πάσχουν από απερίμωση, αλλά ξέρουμε ότι η συγκράτηση των δασών και η δημιουργία νέων δασών μπορεί να καθαρίσει την ατμόσφαιρα. Επομένως είναι ένα μέτρο ήπιας ε, ε, εφαρμογής ε, της κλιματικής αλλαγής. Βεβαίως είναι οικονομικός πλούτος, άρα μπορεί να μας δώσει τη δυνατότητα να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια. Τώρα, γιατί δεν συμβαίνει η δημιουργία δασών με το ρυθμό που θα θέλαμε. Ε, κοιτάξτε, είναι ε, μία περίπλοκη περίπτωση ε, όσον αφορά τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, γιατί μπαίνουμε πλέον σε θέματα χωροταξικά που αφορούν κοινότητες, που αφορούν την εξάπλωση κοινοτήτων. Η κυρία Βάλστρομ έλεγε προηγουμένως ότι έχει αυξηθεί ο πληθυσμός σε επικίνδυνες περιοχές μέχρι και 92% και επομένως μπαίνουμε με την ε, ε, λογική αυτή στα, στα σημεία τα οποία θίξαμε προηγουμένως. Δηλαδή πρέπει να είμαστε σε θέση να πείσουμε τους ε, ηγέτες, αυτούς που είναι υπεύθυνοι για να λαμβάνουν αποφάσεις, να τους πείσουμε για το ορθόνο των σκέψεών μας και βεβαίως να ξεπεράσουμε και προβλήματα προβλήματα που σχετίζονται με την ιδιοκτησία. Γι' αυτό ακριβώς, και έρχομαι στον κύριο Γκέρανς, γι' αυτό είναι σημαντικό ε, να δούμε ποιες ε, μπορεί να είναι οι συμμαχίες που μπορούμε να δημιουργήσουμε με τους ε, υπεύθυνους για την λήψη των αποφάσεων. Εσείς κάνατε συγκεκριμένη ερώτηση για τα τεστ αντοχής των πυρηνικών σταθμών από την αρχή, λόγω και του ρόλου μας ε, όσον αφορά την ε, πρόληψη και αντιμετώπιση καταστροφών, ε, αναμεχθήκαμε, λέω, με τη διαδικασία αυτή. Ο Επίτροπος Ότιγκερ και εγώ η ίδια συζητήσαμε με την, συζητήσαμε πολύ, έχουμε την ομάδα ΕΚΟ η οποία έχει αναμειχθεί πάρα πολύ με τα θέματα αυτά. Ε, διότι τα stress tests είναι πάρα πολύ σημαντικά ε, για τη δουλειά που κάνουμε εμείς ε, Ε, και είναι σημαντικό ε, να καταλάβουν και οι ρυθμιστικές αρχές για την ηλεκτρική ενέργεια και για την ε, πυρηνική ενέργεια και το δικό μας τρόπο σκέψης. Και από την άλλη πλευρά βεβαίως θα πρέπει να γίνονται μελέτες από τις αρμόδιες αρχές τις οποίες θα συμβουλευόμαστε κι εμείς. Αλλά θα ήθελα να διαβρύνω λίγο το θέμα και να πω το εξής. Είναι απολύτως ουσιώδες να έρθουμε σε επαφή με ε, αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις. Ας πούμε, εμείς είχαμε μια ενδιαφέρουσα συνάντηση με τον οικονομικό, ας πούμε, υπεύθυνο της Κομισιόν, τον Επίτροπο Μπαρνιέ, που μπορεί πραγματικά να παίξει πολύ μεγάλο ρόλο ε, στο θέμα της πρόληψης και της αντιμετώπισης ε, των καταστροφών κατά την άποψή μου, μονάχα μέσα από τέτοια συνδυασμένη δράση θα επιτύχουμε. Όχι όταν προσπαθήσουμε εμείς να υψώσουμε τα λάβαρα, ας πούμε, ε, της προσπάθειάς μας. Όχι, όταν συνεργαζόμαστε όλοι. Και όσον αφορά την νομοθεσία στην οποία αναφερθήκατε, ε, κυρία Πρόεδρε, Πρόθεσή μας είναι να ε, δημοσιεύσουμε ανακοινωθέν για την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση ε, καταστροφών ε, κατά προτίμηση φέτος αυτή είναι η φιλοδοξία μου. Γιατί αν θέλουμε να προχωρήσουμε προς τα εμπρός, αν θέλουμε να ενισχύσουμε την δυνατότητα αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών θα πρέπει οπωσδήποτε και το προηγούμενο στάδιο να το καλύψουμε, δηλαδή της ετοιμότητας και της πρόληψης. Θέλω όμως να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Ε, αυξάνεται συνέχεια σε ένταση και σε αυξάνονται συνέχεια σε ένταση και σε ρυθμό και σε συχνότητα οι φυσικές καταστροφές ε, και επομένως προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε ολόκληρο τον κόσμο. Ε, γι' αυτό λοιπόν θα σας ήμουν ευγνώμων εάν εσείς διαρκώς μας πιέζετε για την ετοιμότητα, για την πρόληψη, έτσι ώστε να μην ξεχνάμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα. Το έχω πει πολλές φορές και ίσως έχω κουράσει μερικούς. Τι, αυτό που συνέβη στην Ιαπωνία ήταν πραγματικά κάτι που μου άνοιξε τα μάτια. Τον Μάρτιο του 2011 ε, θα πήγαινα σε μία άσκηση προσωμείωσης σεισμού 5,5, 7,5 ε, αντίστοιχου δηλαδή της, του σεισμού που προκάλεσε το μεγάλο τσουνάμι στην Ινδονησία. Αλλά στην περίπτωση της Φουκοσίμα ξεπεράσαμε κατά πολύ τα 9 μέτρα του κύματος της... Ε, τα εννιά ρίχτερ και το μεγάλο τσουνάμι. Ξεπέρασε η πραγματικότητα και αυτά που είχαμε ε, δει στο παρελθόν. Ευχαριστώ. Θα αρχίσω από τα βάση. Πριν από 20 χρόνια εργαζόμουν στον Ερυθρό Σταυρό και ένα από τα βασικά μας μελήματα ήταν ε, η δεντροφύτευση. Πηγαίναμε παντού και φυτεύαμε δέντρα. Και το θέμα είναι ε, γιατί σταματήσαμε, σταματήσαμε εμείς ε, συνολικά τη γεωργική ανάπτυξη και τη γεωργική εκμετάλλευση. Γιατί έφυγε η γεωργία από τα θέματα της αναπτυξιακής βοήθειας. Αυτά είναι κρίσιμα θέματα και για τις χώρες ε, και για τη διαχείριση του κλιματικού κινδύνου και για τη διατροφική ασφάλεια και την επιστημιστική και για τη μείωση των κινδύνων θεομηνιών. Ως παγκόσμια κοινότητα δεν μπορούμε ε, να κοιτάμε την ευστάθεια και τη σταθερό του πλανήτη μας επειδή είναι της μόδας. Το θέμα με τη διατροφήτευση δεν είναι φιλανθρωπία. Είναι ότι αρχίζουμε να ε, κοιτάμε ε, το θέμα του διοξιδίου του άνθρακα και τη διαχείριση του που είναι ένα πολύ δαπανηρό ζήτημα και θεωρούμε πλέον ε, το δάσος πραγματικό κεφάλαιο για χώρες όπως είναι το Νεπάλ, ε, για παράδειγμα, που έχει μπει στο πρόγραμμα, έχουν μια πολύ μεγάλη δυνατότητα, ένα ενεργητικό, ένα ατού που μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Και είδαμε ότι έχουμε φαινόμενα κατολιστήσεων και σαρωτικών πλημμυρών σε αστικές περιοχές και συνδέονται αυτά με τα δάση και τα δέντρα πού φτάνει στα όρια της η πρόληψη και τι μας έκανε να συνειδητοποιήσουμε η Φουκουσίμα. Για μένα ε, το κρισιμότερο βέβαια και το συζήτησα με συναδέλφου στην Ιαπωνία είναι το εξή. Ο κάθετος ε, κατακόρυφος τρόπος με τον οποίο ε, διοικούμε τις χώρες μας. Ποιος αποφασίζει ε, τα επίπεδα κινδύνου. Ούτε ο ιδιωτικός τομέας, ούτε οι μηχανικοί που σχεδιάζουν ε, τα εργοστάσια και ούτε οι ιδιώτες που πληρώνουν αυτές τις επενδύσεις. Σήμερα κανένας ιδιώτης δεν επενδύει ε, σε πυρηνικά εργοστάσια, μόνο τα κράτη, γιατί είναι πάρα πολύ δαπανηρή αυτή η επένδυση. Λοιπόν, ποιος αποφασίζει για τα επίπεδα κινδύνου. Για τελικά και οι κυβερνήσεις και οι ιδιώτες θα πληρώσουν τις ε, ζημίες της ε, αισιόδοξη ε, βαφή σχεδιασμού. Λοιπόν, για πρώτη φορά διεθνώς καταφέραμε να συναντήσουμε μια επιτροπή που ασχολείται με τις πυρηνικές εκρήξεις και για μη πολεμικούς σκοπούς και τέτοιου είδους φαινόμενα, ας πούμε, πυρηνικά εργοστάσια που ασχολούνται και με ε, σεισμούς και, ε, και άλλα πυρηνικά ατυχήματα και άλλα ατυχήματα. Όλα αυτά ποιος τα διαχειρίζεται σε διαφορετικά επίπεδα ή εμπειρογνώμονες, καλώς, αλλά συνολική ε, θεώρηση υπάρχει, συνολικοί μηχανισμοί ολοκληρωμένοι και διεθνείς και σε επίπεδο κρατών. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ το έχει θέσει αυτό το θέμα και μάλιστα τάραξε τα νερά. Ζήτησε ε, από το σύστημα οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών να ε, κάνουμε μια αναφορά, μια συλλογή στοιχείων για το πώς συνεργαζόμαστε και θα έχουμε το Σεπτέμβριο ε, κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών μια ευρύτατη συζήτηση σε πολύ ψηλό επίπεδο. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί συζητούμε για όλους τους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας πληθυσμός σε καιρό ειρήνης Και θα πρέπει λίγο να συνεργαστούμε, να χαλαρώσουμε τις άμυνες του καθένα και να το δούμε σφαιρικά και συνολικά. Πώς ορίζεται ο κίνδυνος. Τι εστί κίνδυνος. Ε, πολύ συχνά είναι τοπικός, αν και γίνεται μεγάλος λόγος σήμερα για παγκόσμιους κινδύνους. Αλλά υπάρχουν και στάνταρ εκεί, υπάρχουν περιφερειακοί κίνδυνοι, εθνικοί, τοπικοί και αλλάζει αυτό. Και κλασικό παράδειγμα είναι η κλιματική αλλαγή, ε, είναι ε, μετρολογικά φαινόμενα, τα ποτάμια αλλάζουν συμπεριφορά. Κάποια φράγματα, όπως είδαμε στις Ηνωμένε Πολιτείε που έχουν ε, κατασκευαστεί πριν από 30 χρόνια, σήμερα αποδεικνύονται ανίσχυρα και κοιτάξτε τι έγινε στον Ινδό ποταμό στο Πακιστάν. Χρειάζεται λοιπόν μια συνεχής εκτίμηση κινδύνου και ε, μάλιστα να διατίθεται δωρεάν αυτή η πληροφόρηση στους πολίτες, γιατί και οι ευθύνε είναι και των πολιτών, ξέρετε. Εμείς ως μεμονωμένοι πολίτες δεν μπορούμε να τα περιμένουμε πάντα από την πολιτεία, από την κοινωνία των πολιτών. Είναι προσωπικό ζήτημα του καθενός, ατομική ευθύνη. Και όταν ε, είναι κανείς καλά ενημερωμένος, κάνει και τη δουλειά του. Καθαρίζει, ας πούμε, τους υπονόμους που βρίσκονται στη ε, γειτονιά του για να μην πλημμυρίσει το υπόγειο του σπιτιού του. Από εκεί ξεκινάει η προσπάθεια αυτή. Yep, okay. um... Θα αρχίσω κι εγώ με τα δέντρα που έχει ενδιαφέρον η ιστορία αυτή. Εξετάστε τις πλημμύρες που έγιναν ε, πέρσι στο Πακιστάν και πλήγησαν 20 εκατομμύρια άνθρωποι από τις χειρότερες πλημμύρες που έχουμε δει στους σύγχρονους καιρούς. Εάν εξετάσετε τώρα τις κοιλάδες αυτές, κίτες μάλλον των ποταμών, αν τις εξετάσετε τις κίτες των ποταμών ως οικολογικό σύστημα, θα δείτε ότι αυτό που συνέβη είναι ότι υπήρξε σε τεράστιο βαθμό αποψήλωση δασών στις περιφερειακές ε, περιοχές γύρω από τα ποτάμια, αυτό που γίνεται όταν κόψετε τα δέντρα είναι ότι η απορροφητικότητα του εδάφους σε νερό μειώνεται. Επομένως, αρχίζετε να αυξάνεται έτσι τους όγκους νερού που θα καταλήξουν τελικά στο ποτάμιο σύστημα, αυξάνεται και η ταχύτητα του νερού, άρα διαβρώνει τα εδάφη περισσότερο άρα μεταφέρει και περισσότερο ίζημα, καταβαίνει λοιπόν περισσότερο ίζημα, ε, κατεβαίνει με μεγαλύτερη ταχύτητα σε μεγαλύτερες ποσότητες και στα κατάντη των ποταμών έχουμε ε, φτιάξει φράγματα, συστήματα ε, οδών, έχουμε κανάλια για την απομάκρυνση των νερών Οποιαδήποτε λοιπόν ικανότητα που είχε δημιουργηθεί πριν όταν ερχόντουσαν οι μουσώνες ε, έχει τώρα καταστραφεί. Δηλαδή έχουμε βάλει ένα είδος ζουρλομανδία. Έχουμε αυξήσει τις ίσροες ενώ ταυτόχρονα έχουμε περιορίσει τις έκροες, τις δυνατότητες έκροης στο έβγα του ποταμού. Ήταν λοιπόν πραγματικά μαθηματικός βέβαιον ότι θα γίνουν οι πλημμύρες αυτές σε περιόδους μουσώνων. Σε περιόδους μουσώνων. Και το πιθανόν είναι ότι ε, θα ξαναγίνει και ακόμα χειρότερα. Διότι το πρόβλημα είναι ότι έχουμε επηρεάσει με τέτοιο τρόπο το περιβάλλον, ώστε δεν αντιποκρίνεται πλέον στην, ε, ανάγκες της φύσης. Ο Σουμάκερ που ήταν ε, παλιός μελετητής ε, της δεκαετίας του 60 ε, είχε γράψει ένα βιβλίο που το έλεγε Small is Beautiful και που έλεγε ότι η παρέμβαση του ανθρώπου δηλαδή πρέπει να είναι περιορισμένη. Αυτό που κάνουν τα φυσικά οικοσυστήματα είναι ότι έχουν ένα ρόλο ρυθμιστικό των ακραίων φαινομένων. Δηλαδή, δηλαδή μπορούν να απορροφήσουν τα ύδατα, μπορούν να τα κάνουν, να εκρέψουν με τρόπο ακίνδυνο, αλλά αυτό που έχουμε κάνει στην πραγματικότητα είναι ότι έχουμε παρεμβάλει ένα οικονομικό σύστημα το οποίο δεν αξιολογεί ή δεν ε, αξιοποιεί τις υπηρεσίες που προσφέρουν τα οικολογικά συστήματα. Ήταν η αξία του ξύλου που το κόψαμε και το μεταφέραμε στις αγορές. Ενώ ε, ε, οι υπηρεσίες που πρόσφεραν τα δέντρα, τη συγκράτηση των νερών, του καθαρισμού των νερών που τελικά κατέληγαν στο, έδαφο, στο, στο έδαφος κτλ. Αυτά αγνοήθηκαν. Υπάρχει δυνατότητα τώρα, εάν χρησιμοποιήσουμε το Red Reforestation Funding, το οποίο είναι ένα ταμείο, μια χρηματοδότηση για την μείωση του διοξιδίου του άνθρακος, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να ε, προσαρμόσουμε τις ικανότητες των ε, συστημάτων στα ανάντι των ποταμών, δημιουργώντας ή ενισχύοντας πάλι έτσι τις ικανότητες των οικοσυστημάτων να απορροφήσουν τα ακραία φαινόμενα και να μειώσουν έτσι τους κινδύνους για τους πληθυσμούς που βρίσκονται στα κατάντι των ποταμών. Άρα, αυτά όχι μόνο αυξάνουν την ικανότητα του φυσικού περιβάλλοντο, δημιουργούν και απασχόληση, μειώνουν και του κινδύνου. Αυτά λοιπόν μπορούν να ενισχυθούν εάν φερθούμε με ευφυή τρόπο για τι επενδύσει που θα κάνουμε. Και βέβαια, να βάλουμε και τους ντόπιου μέσα στη διαδικασία αυτή. Διότι μόνο εάν οι τελικοί χρήστες ε, τελικά των υπηρεσιών αυτών ε, συμμετάσχουν και στατευθούν και αυτοί, τότε θα αποδώσει το σύστημα. Και βεβαίως η αντίληψη που έχει το κοινό για αυτά είναι απόλυτα κρίσιμη. Η, αντίληψη του κοινού στο Πακιστάν πιθανώς θα έχει αλλάξει τώρα μετά από αυτές τις ε, ακραίες πλημμύρες η αντίληψη του κοινού, των Ιαπώνων δηλαδή, για την ασφάλεια ε, των πυρηνικών εγκαταστάσεων της ανατολικής ακτής τους θα έχει αλλάξει φαντάζομαι ραγδαία μετά από τα ε, πυρηνικά αυτά ατυχήματα. Επομένως, η αντίληψη του κοινού, η συνειδητοποίηση από πλευράς κοινού είναι απόλυτα απαραίτητη για να ε, δημιουργηθεί η εντύπωση για το πού βρίσκεται αυτό το ακραίο κατόφλι το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνεται. Βεβαίω θα ζούμε πάντα με τον κίνδυνο. Το ζήτημα είναι πώς περιορίζουμε τον κίνδυνο σε αποδεκτά επίπεδα και πού κάνουμε τις ανταλλαγές, τα trade-off. Ανάμεσα δηλαδή στην ταχεία οικονομική ανάπτυξη και στην αυξημένη ε, έκθεση σε κινδύνους, το ευάλωτό μας απέναντι στους κινδύνους. Ας μπουν λοιπόν και οι πολίτες των τοπικών κοινωνιών στην πολιτική διαδικασία, γιατί αυτό θα εξασφαλίσει μια πολύ πιο εξισορροπημένη προσέγγιση εν τέλει. Η πρόεδρος κυρία Στρίφλερ, ευχαριστώ. Τρεις ερωτήσεις ακόμη. Και πρώτα, ο κύριος Κασμανιάκ. Ευχαριστώ πολύ κύρια Πρόεδρε και ευχαριστούμε πάρα πολύ τους καλεσμένους μας για τους, ε, για τις εξαιρετικές ομιλίες τους. Ακούω και ξανακούω αυτά που λέγονται και κατανοώ ότι τελικά το ποιος, η λέξη κλειδί είναι συνειδητοποίηση. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν όλοι πώς έχουν τα πράγματα. Δεν θέλω να είμαι ε, ηρωνικός, αλλά πάντως έχω την εντύπωση, γιατί αυτή η ηρωνία τρέφεται και εναντίον μου, έχω την εντύπωση ότι κάποιοι... Ε, πολιτικοί ε, σαν να χαίρονται σε φυσικές καταστροφές γιατί ανασκουμπώνουν τα μανίκια τους και ε, πηγαίνουν ε, στα μέρη έτσι που έχουν πληγή και επομένως αυτή η φυσική καταστροφή γίνεται ένα μέσο επικοινωνίας για να δείξουν ότι μπορούν να πετάξουν και τη γραβάτα και το σακάκι και γίνεται κατά κάποιο τρόπο πολιτική επένδυση μέσα από αυτές τις ε, φυσικές ε, ε, καταστροφές. Απ' την άλλη πλευρά διαπιστώνω ότι υπάρχει μία τάση, ακόμα και οι φυσικές καταστροφές, να θεωρούνται επενδύσεις. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Οι επενδύσεις πρέπει να γίνουν πριν από τις φυσικές καταστροφές, πριν γίνουν οι, οι πλημμύρες. και ε, από την άλλη πλευρά μας λένε, ακούμε πολύ συχνά, θα κάνουμε ένα σωρό επενδύσεις ε, και τελικά οι επενδύσεις αυτές δεν θα επιστρέψουν χρήματα αφού δεν θα γίνουν ποτέ καταστροφές ή δεν θα γίνει ποτέ ε, κάποια πλημμύρα. Διευθυντικά ταμεία, κυρία Επίτροπε, ε, που όπως είπατε και εσείς οι ίδια παρουσιάζουν πολύ μικρό επίπεδο ε, απορρόφησης. Ε, γιατί αυτό οι περιφερειακές αρχές, οι τοπικές αρχές δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν τα χρήματα αυτά. Μήπως προτιμούν, επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν διαφορετικά τα χρήματα. Ευχαριστώ πολύ, Κέλλερ. Ευχαριστώ. Ως πράσινη χαίρομαι πάρα πολύ που όλοι μιλούν για δεντροφύτευση αυτή τη στιγμή και συμφωνώ και χαίρομαι που όλοι συμφωνούν. Πολύ ωραία ιδέα. Ανέκαθεν άλλωστε και είναι κρίμα που δεν το είχαν εκτιμήσει στο παρελθόν όσο χρειαζόταν και δεν μας άκουγαν όταν τα λέγαμε εμείς αυτά. Σας ευχαριστώ για τις ε, εισηγήσεις σας και βεβαίως θεωρώ πάντα ότι η πρόληψη είναι καλύτερη από την αντιμετώπιση, αλλά καλό είναι να έχουμε και ένα περιθώριο για την αντιμετώπιση. Πολλές είναι οι περιπτώσεις που δείχνουν ότι μπορεί κανείς να κάνει πάρα πολλά από την πρόληψη. Ε, ακούσαμε για τη Χιλία, αλλά και το Μπαγκλαντές, που έχει πέσει σημαντικά ο ρυθμός των θανάτων με πολύ λίγα και εύκολα μέτρα πρόληψης, ε, αντιμετώπιση των πλημμυρών, ας πούμε, που είναι πολύ συχνές και επαναλαμβανόμενες. Βέβαια, μου έχει προκαλέσει και λίγη κατάθλιψη και μελαγχολία αυτές τις συζητήσεις, γιατί τα λέμε ξανά και ξανά και εδώ στην Επιτροπή μας δεν είναι η πρώτη φορά. Όλο τα ίδια λέμε και βασικά όλοι γνωρίζουμε τι χρειάζεται να γίνει. Είναι απλή δουλειά. καλύτερη ε, αντισυσμική ε, ε, κατασκευή των κτηρίων, καταπολέμηση των πλημμυρών. Όλοι γνωρίζουμε τι σημαίνει αύξηση τη συνειδητοποίηση και ότι δεν μπορεί να επιβληθεί άνωθεν. Όλα αυτά τα γνωρίζουμε πολύ καλά, αλλά δεν συμβαίνουν ακόμα σε πολλέ χώρε και σε πλούσιε όπω οι Ηνωμένε Πολιτείε. Κάθε χρόνο έχουν του ίδιου άνεμος και κυκλώνε και τέτοια στι ίδιε περιοχέ, αλλά κάθε χρόνο είναι τρομερή θεομηνία και λένε «Ω Θεέ μου πάλι έρχεται» το κλίμα χειροτερεύει παντού στον κόσμο και βλέπουμε τι γίνεται με την κλιματική αλλαγή. Είναι πιο ακραία τα καιρικά φαινόμενα πλέον. Αλλά όλα αυτά δεν τα βλέπω και αυτή τη συνειδητοποίηση που πρεσβεύετε κι εσείς και όλοι επαγγελόμαστε. Δεν βλέπω να μεταφράζεται σε πολιτική βούληση, τουλάχιστον όχι παντού και εν πάση περιπτώσει όχι σε περιοχές που την έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη. Δεν ξέρω, εντάξει, τα μικρά βήματα τα κάνετε κι εσείς και, και στην Ευρώπη κάνουμε διασκέψεις και συζητάμε, ωραία αυτά. Αλλά φαίνεται ότι δεν φτάνουν στον προορισμό τους αυτά και δεν καταλαβαίνω γιατί. Γιατί μέχρι τώρα όλοι έχουν συνειδητοποιήσει ότι είναι πολύ ακριβή αυτή η ιστορία, όλοι έχουν συνειδητοποιήσει ότι κοστίζει και πολλέ ψήφου. Γιατί όμω ο κόσμο δεν αντιδρά, τι τον σταματά, τι τον κάνει, δεν ξέρω. Από τη μια Μπορεί κανείς να πει ε, ότι δεν έχουμε πλημμύρες τα τελευταία 20 χρόνια και γιατί να έχουμε τώρα. Αλλά κάποιοι άλλοι γνωρίζουν ότι θα γίνουν ε, αυτές οι πλημμύρες, ότι θα έρθει το φυσικό φαινόμενο και πάλι δεν κάνουν τίποτα. Εσείς που τους συναντάτε και συζητάτε πώς το εκτιμάτε, τι πρόβλημα έχουν και δεν μπορούν να εφαρμόσουν αυτά που λέμε. Και μετά ε, κάτι προς την κυρία Γεωργίευα που μιλήσετε για ρεσιμότητα, δηλαδή βάλουμε όρους ε, για τις ε, εκροές ε, έτσι, αναπτυξιακής βοήθειας να μειώνει το κίνδυνο ή να υπάρχει θέμα πρόληψης των θεομηνιών. Και πώς θα γίνει αυτό, πώς το φαντάζεστε, γιατί τελικά πότε θα βοηθήσουμε αυτούς που το έχουν ανάγκη. Αυτό θα πρέπει να κάνουμε. Και είναι προφανές και ανεφόρον, γιατί όρος για ποιο πράγμα. Γενικά δεν με πείθει αυτό το θέμα της ερεσιμότητας ότι θα βοηθήσει και θα βελτιώσει τα πράγματα. Πάντως περιμένω να ακούσω και τις δικές σας απαντήσεις. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κάσμαν. Um, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εκφράζω τη λύπη μου που δεν ήμουν παρόν από την αρχή της συζητήσεως. Πάντως ε, άκουσα με εξαιρετικό ενδιαφέρον τα όσα ελέγχθηκαν. Βεβαίω, στον πραγματικό κόσμο υπάρχουν έντονες πολιτικές πιέσεις για τις δωρήτριε χώρες να αναλάβουν, μάλλον να ε, εκπληρώσουν ε, δεσμεύσεις, υποσχέσει τις οποίες είχαν αναλάβει τους καιρού που ήταν τα πράγματα οικονομικά καλά. Η ανάπτυξη είναι στην ουσία επένδυση και στις δικές μας ζωές, ε, διότι επενδύουμε στις ζωές των άλλων και συμφωνώ απόλυτα εδώ με τον κύριο Όξλε και με τα όσα εξήγησε ότι δηλαδή πρέπει να γίνει στο τοπικό επίπεδο, πρέπει να δώσουμε δύναμη στους ανθρώπους εκείνους. Πρέπει να τους προσφέρουμε τη δυνατότητα να αναπτύξουν ικανότητες στο τοπικό επίπεδο, γιατί αλλιώς όποιες στρατηγικές και να επιλέξουμε, ποτέ δεν θα μπορέσουμε να προλάβουμε, να επιτύχουμε δηλαδή τις προληπτικές εκείνες δράσεις που πρέπει να γίνουν επιτόπου. Δεν θυμούμε πώς λεγόταν ε, το πρόσωπο εκείνο όταν είχαμε πάει τον Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη σε μια συνάντηση NDG, ένας ε, πραγματικά λαμπρός εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών, μας είχε απευθύνει σύντομη ομιλία για τη λεγόμενη connectivity, την διασύνδεση των πάντων. Και αυτό είναι που πρέπει να επαναφέρουμε ως στοιχείο στον πολιτικό μας διάλογο, ε, στην πολιτική μας στις πολιτικές μας θέσεις. Διότι αυτά που συμβαίνουν στην άλλη άκρη του κόσμου, για παράδειγμα στην Ιαπωνία, επηρεάζουν ολόκληρο τον πλανήτη. Η προσέγγιση, για παράδειγμα, για την συνοχή. Θα, θα χρειαστεί να έχουμε συνοχή σε όλες μας τις πολιτικές και σε όλες τις προσεγγίσεις για την επίλυση των προβλημάτων. Δεν θα επιτύχουμε τίποτε χωρίς χρήματα. Τα χρήματα είναι αυτά, το χρήμα είναι αυτό που θα δώσει τις δυνατότητες, διότι δίνει και πληροφορίες και ενημέρωση δηλαδή και τη λεγόμενη ownership, δηλαδή το να νιώσουν οι άνθρωποι ότι είναι κύριοι της διαδικασίας. Πιο, ε, σημαντική, ενισχυμένη ε, ανταπόκριση στην, ε, στο παγκόσμιο επίπεδο, ανταπόκριση στις φυσικές καταστροφές ε, παρεμπόδιση παράνομη αλληλεία ούτω καθεξή. Όλα αυτά είναι η διαφύλαξη των κοινών αγαθών. Όλα αυτά είναι ωραία. Υπέροχα. Αλλά αυτό που θέλω εγώ ε, να εξασφαλίσω είναι ότι θα πέσουν σε καρποφόρο έδαφο, ότι θα υπάρχει νερό ώστε το δενδράκι να μπορέσει να αναπτυχθεί. Αυτή λοιπόν είναι η ολιστική ε, προσέγγιση που οφείλουμε να επιλέξουμε. Βεβαίω και υπάρχει αντίληψη του κοινού όταν έχουμε για παράδειγμα τρομερές οικολογικές καταστροφές όπως στην Αϊτή, όπως στην Ιαπωνία. Αλλά αυτά γίνονται εδώ και αιώνες. Και η αντίληψη του κοινού βεβαίως ε, ε, υφίσταται και την λύθη και την ελπίδα ότι δεν θα ξανασυμβεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Επίτροπο μάλλον, με γνωρίζει, με έχει ξανακούσει πολλέ φορέ και γνωρίζει περίπου τι λέω. Αλλά πολιτικά στην ουσία είμαστε εσωστρεφείς αυτό που πρέπει να γίνει είναι να συνεργαστούμε, να ξεφύγουμε από αυτή την εσωστρέφεια, την καταθλιπτική εσωστρέφεια, η οποία δεν αποδίδει τίποτα. Διότι εν τέλει οι έξωθοι επιβαλλόμενες λύσεις για τις ε, θεομηνίες και άλλες καταστροφές είναι πάντοτε second best και τελικά δεν αποδίδουν αυτό που θα έπρεπε. Και θα δώσω το, ρολ, λόγο. Ποιος θα ξεκινήσει, θα ξεκινήσουμε ανάποδα. Uh, Θα ξεκινήσουμε ανάποδα λοιπόν από τον κύριο Όξλεϊ. Ξέρετε, αυτό το ζήτημα των καταστροφών το λέμε, το ξαναλέμε. Νομίζω ότι η καλύτερη ευκαιρία για να προχωρήσουμε το θέμα αυτό της πρόληψης των κινδύνων είναι ακριβώς μετά από μια μεγάλη καταστροφή γιατί αλλάζει ο τρόπος, η οπτική γωνία του κοινού, ο κόσμος βλέπει διαφορετικά τα πράγματα εκείνη την ώρα που ο αντίκτυπος ακόμα είναι μεγάλος. Ε, ε, είναι, υπάρχουν ε, οι ανθρωπιστικές αρχές οι οποίες πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα κτλ. Νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό μπορεί κανείς να εξηγήσει καλύτερα το θέμα ε, της ε, πρόληψης και δεν νομίζω ότι χρησιμοποιούμε και ε, ότι πραγματικά δρατόμαστε των ευκαιριών που δίνουν αυτές οι καταστροφές. Και βεβαίως θα πρέπει με συστημικό τρόπο να δούμε γιατί συμβαίνουν συχνά οι καταστροφές στο Πακιστάνι, γιατί γίνονται οι καταστροφές και τι είδους είναι αυτές που λαμβάνουν χώρο στην Ιαπωνία ας πούμε πάντα ε, ε, δεν κάνουμε ποτέ ε, μία post-mortem ανάλυση της κατάστασης και αυτό νομίζω ότι αποτελεί έλλειψη στο σύστημα. Θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε μία έρευνα τύπου μαύρου κουτιού αεροπλάνου να, να, να, ανοίξουμε το μαύρο κουτί, να το βρούμε, να το διαβάσουμε για να καταλάβουμε ποιες είναι οι ανεπάρκειες, ποιες είναι ε, οι ελλείψεις ε, των ε, διαδικασιών που ακολουθούμε. Μαθαίνουμε, πρέπει να μαθαίνουμε από τις καταστροφές και να ανοίξουμε την ευκαιρία που μας δίνεται, την πολιτική ευκαιρία κιόλας μετά από τέτοιες καταστροφές έτσι ώστε να αποφευχθούν στο μέλλον παρόμοιες καταστροφές. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει ε, να αναγνωστεί συγγένεια ανάμεσα στην πρόληψη, το ατύχημα ε, ε, και δεν θέλω να πω τίποτα άλλο γι' αυτό. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να σας ενθαρρύνω λίγο και να σας πω ότι τα πράγματα έχουν αρχίσει και κινούνται. Συμφωνώ μαζί σας ότι όταν μαζευόμαστε τίνουμε να επαναλαμβάνουμε ποια είναι τα εμπόδια, ποιες είναι οι δυσκολίες. Ε, ακούσαμε για το Πακιστάν, για τον Μπαγκλαντές, αλλά εγώ μπορώ να σας αναφέρω την περίπτωση της Κίνας με μεγάλη ανάπτυξη. Τώρα που έχουν λίγο σταθεροποιηθεί στο ρυθμό της ανάπτυξης τους, αρχίζουν και αντιμετωπίζουν κάποια έτσι πιο λεπτά ζητήματα. Και και ακόμα και οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν ας πούμε κάποιες οικιστικές, ε, ε, κάποιες ε, χωροταξικές επιλογές που έχουν αναλάβει και προκρίνει, οι οποίες αναγνωρίζεται ότι θα δημιουργήσουν προβλήματα στο μέλλον. Ήδη η αναγνώριση αυτή είναι τεράστια ε, πρόοδος κατά την άποψή μου. Στην Αυστραλία επίσης ε, υπάρχει ένα μεγάλο ε, πρόγραμμα για τις φυσικές καταστροφές, National Resilience Plan, Πιστεύουμε ότι τα απλά προγράμματα, αυτά τα οποία ε, δημιουργούν ε, ε, άμεσα κίνητρα, αυτά τα οποία έχουν σαν προϋπόθεση την αιρεσιμότητα, ενδεχομένως να είναι πιο περίπλοκα. Πρόσφατα είχα μία συνάντηση με εκπροσώπους ασιατικών χωρών, και ανέφερα την αρχή της αιρεσιμότητας, αλλά μου είπαν ότι ξέρετε σε εθνικό επίπεδο, σε διεθνές επίπεδο μπορεί να είναι δημοφιλής αυτή η ιδέα, αλλά όχι σε ε, διεθνές, όχι σε εθνικό. Ε, ανέφερα την ε, περίπτωση του Περού. Εκεί ο πρόεδρος Γκαρσία κατάλαβε ότι δεν θα μπορούσαν μέσω των απλών γραφειοκρατικών, συνήθων γραφειοκρατικών ε, διαδικασιών να ξεκινήσουν την δενδροφύτευση ε, με, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές. Όμως ε, είπε στον Υπουργό των Οικονομικών ότι εάν κάνουν σωστά προγράμματα πρόληψης τότε θα απελευθερωθούν κονδύλια. Ε, και μάλιστα το Υπουργείο βοήθησε με τεχνογνωσία, με πραγματογνωμοσύνη ε, και πραγματικά νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε τέτοιες δράσεις. Νομίζω ότι το σημαντικό στοιχείο είναι να έχουμε καλή αντίληψη της ε, κατάστασης. Διαπιστώνουμε ότι ε, δίνουμε υπερβολική προβολή στις μεγάλες ε, καταστροφές, αλλά λίγο σαν ε, γεγονότα μόνο. Εμείς προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε τους δημοσιογράφους έτσι ώστε να παρουσιάζουν τις καταστροφές με τρόπο ώστε να εκπαιδεύουν και τον κόσμο κατά κάποιο τρόπο. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε επίσης ε, συνεκτική όταν αντιμετωπίζουμε το, θέμα της πρόληψης και της αντιμετώπισης και βεβαίως καταλαβαίνω ότι έχουμε την βιώσιμη ανάπτυξη, έχουμε την ανάπτυξη, έχουμε ε, τους, τα χρηματοπιστωτικά ε, ιδρύματα. Βεβαίως είναι ένα περίπλοκο ζήτημα, αλλά πιστεύω ότι θα το λύσουμε μόνο εάν όλοι μαζί σε ένα κοινό πρόγραμμα, σε, με προσπάθειες συντονιστούμε ε, σε ένα κοινό πρόγραμμα. Ελλείψεις υπάρχουν. Ε, και δεν είναι ότι δεν υπάρχουν παράλληλες πορείες, είναι ότι η αρμή ανάμεσα σε αυτές τις παράλληλες τροχιές δεν κρατάνε καλά. Η συγκολητική ουσία δηλαδή δεν ε, είναι καλή. Πάντως πιστεύω ότι βλέπω και διαπιστώνω ότι πολλές κυβερνήσεις, ε, πολλέ, πολλοί πολυμερείς οργανισμοί και πολυμερεί ιδρύματα προσπαθούν ε, να αντιμετωπίσουν ε, τέτοια ζητήματα έτσι από κοινού. Διαπιστώνω επίσης ότι σε πολλές περιπτώσεις έχουμε υψηλού επίπεδου πολιτική δέσμευση και το σημαντικό είναι πώς μπορούν να διατεθούν κονδύλια σε τοπικές ε, κυβερνήσεις για τοπική δράση. Επίσης πώς μπορούμε να συντονίσουμε ε, την ε, δράση των, ε, ε, των δωρητών, ε, γιατί οι δωρητές και κάποιοι φορείς έτσι, που δίνουν χρήματα έχουν την τάση να είναι και λίγο παρεμβατικοί στον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστεί το θέμα. Νομίζω ότι ο καθένας προσπαθεί να βρει ένα τρόπο ε, να επιταχύνει την διαδικασία και να δώσει περισσότερες αρμοδιότητες στις τοπικές κυβερνήσεις. Κύριε ε, Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Κάσμαρεκ ε, είπε κάτι πάρα πολύ σωστό. Η αντιμετώπιση των ε, καταστροφών, των μεγάλων καταστροφών, είναι στα μεγάλα δελτία ειδήσεων. Ε, τα προληπτικά μέτρα ποτέ. Γι' αυτό ε, δεν μπορεί να είναι πολύ μεγάλη προτεραιότητα η πρόληψη. Αλλά δεν είναι αυτός μόνο ο κυριότερος λόγος. Γιατί αυτή τη στιγμή έχει επιβραδυνθεί λίγο η απορρόφηση των κονδυλίων ε, για τους κινδύνους των θεομηνιών. Κύριος, αυτό που συμβαίνει για τις πλημμύρες ας πούμε, για τη βελτίωση της υποδομής. Είναι έργα πάρα πολύ περίπλοκα. Ε, πολλές φορές χρησιμοποιούν πολλούς κλάδους από τις υποδομές, τη γεωργία, την αστική ανάπτυξη, την ανάπτυξη της υπαίθρου. Πολλές φορές χρειάζονται πάρα πολύ περίπλοκα σχέδια τα οποία συγκρούονται με τα συμφέροντα διαφόρων ε, κοινοτήτων και δεν είναι ένα παιχνίδι από που κερδίζουν όλοι. Ορισμένοι κερδίζουν, άλλοι πάλι χάνουν. Γι' αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο να στηθούν αυτά τα προληπτικά μέτρα. Είναι πιο εύκολο να φτιάξει, α πούμε, ένα αυτοκινητόδρομο με υποστήριξη των διαρθρωτικών ταμείων. Αλλά γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να εργαστούμε σε αυτή την κατεύθυνση και να καταλάβουμε τη φύση τη πρόληψη. Ότι είναι πολλοί κλάδοι που συνδέονται θα πρέπει να συνεργάζονται πολύ και εμείς ε, με θεσμικούς ε, φορείς που ασχολούνται με το περιβάλλον ή και τις τοπικές κοινότητες, γιατί πολλές φορές αντιδρούν οι κάτοικοι. Γιατί λένε, ωραία, εντάξει, είναι κακό, είναι θεομηνία. Αλλά άμα μου απολωτριώσεις ε, το χωράφι μου και χάσω το εισόδημά μου, τι να το κάνω και δεν έχω και δρόμο. Ε, και πραγματικά δεν είναι καθόλου αυκαταφρόνητο το να κάνουμε τοπικό πληθυσμό να το καταλάβει και να είναι προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω. Συμφωνώ απολύτως με τη Μαργαρέτα για το θέμα του αυτό. Το ποτήρι είναι μισό γεμάτο, δεν είναι μισό άδειο. Τα πράγματα έχουν κινηθεί. Η Κωνσταντίνα, για παράδειγμα, είναι μια χώρα όπου είναι πραγματικότητα οι πληρωμές για οικολογικές υπηρεσίες. Δηλαδή ένα δέντρο παράγει νερό, δεσμεύει διοξίδιο του άνθρακα και φέρνει εισόδημα ε, σε ένα κάτοικο. Οπότε αν το κόψει αυτό το δέντρο χάνει. Και άλλα παραδείγματα μπορούμε να φέρουμε, αλλά δεν έχει έρθει ακόμα αυτή η κρίσιμη μάζα που θα αλλάξει τα πράγματα. Για ποιο λόγο. Απαντώ στον κύριο Κασμάρεκ ότι... Ε, και πάλι λέγοντας ότι από τη φύση της η πρόληψη συνδέεται με πολλούς τομείς και μπαίνουν στη μέση συμφέροντα. Κοιτάξτε το Πακιστάν που συζητήσαμε προηγουμένως. Αν θέλει κάποιος να αντιμετωπίσει διορθωτικά αυτό το πρόβλημα επί σειρά ετών, τι σημαίνει. Ότι θα πρέπει να διώξουμε κόσμο ε, σε ένα πολύ πυκνοκατοικημένο κομμάτι της χώρας που κατοικούν εκεί και πολιτικές που να αλλάξουν πάρα πολύ τη χρήση της γης ε, με, με κίνητρα ε, που τους εγκατέστησαν τα κίνητρα για την εκμετάλλευση της γης εκεί. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι συνδυασμό οικονομικών συμφερόντων, ακριβώ η πρόληψη δεν είναι στα δελτία των ειδήσεων στην τηλεόραση. Γι' αυτό είναι και τόσο δύσκολο. Αλλά και γι' αυτό θα πρέπει να το συζητούμε και να προωθούμε την υπόθεση αυτή βήμα-βήμα. Για το θέμα της αιρεσιμότητας. Είναι δύο ειδών η μία συνδέεται με τον αναπτυσσόμενο κόσμο και δεν αφορά τόσο πολύ τις κυβερνήσεις, αλλά και την κοινότητα των εργαζομένων σε θέματα αναπτυσσιακά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι πολύ απλό αυτό το βήμα και μπορεί να γίνει. Σας ε, μίλησα για τα προφίλ και την περιγραφή 31 ε, χωρών που είναι οι χώρες εκείνες που απειλούνται περισσότερο από τις θεομηνίες. Να καταλάβουμε τους κινδύνους και όταν υποστηρίζουμε κάποια προγράμματα να είναι εκείνα τα προγράμματα που θα ενισχύσουν την αντοχή ε, των χωρών αυτών και δεν θα την αποδυναμώσουν. Γι' αυτό είναι εκ των όνου κάνευ για την ε, αναπτυξιακή βοήθεια. Θέλουμε να είμαστε ουσιαστικοί εταίροι και να βοηθούμε τις χώρες αυτές. και να ξέρουμε ότι είναι μακρύς ο δρόμος. Στην Κίνα, εγώ είχα εργαστεί σε ένα πρόγραμμα, ε, σε ένα ε, οροπέδιο έτσι, ε, με γη λος αργυλώδη που ήταν πάρα πολύ κατεστραμμένο και αυτό το πρόγραμμα έχει διάρκεια τουλάχιστον 25 ετή ίσως και περισσότερο. Και από εκεί και πέρα αρχίζεις να βλέπεις τα αποτελέσματα, αλλά δεν θα πρέπει να χαλαρώνουμε ε, στις προσπάθειες. Δεν τροφιτεύαμε χρόνο, το χρόνο για να αλλάξει το οικοσύστημα και να αλλάξει η γη. Σήμερα είναι τελείως διαφορετική εικόνα από ό,τι πριν από 15 χρόνια και το πρόγραμμα ε, συνεχίζει να τρέχει. Και αν μου επιτρέπετε να τελειώσω με την Κίνα και πάλι, γιατί αναφέρετε κι εσείς το 2,7% του ΑΕΠ. Στη δεκαετία του 90 είχα το τεράστιο προνόμιο να συνεργάζομαι με την Κίνα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα χώρα αυτή για όλους και για από πάση ε, σε θέματα. Λοιπόν, η ε, Κίνα ε, φιλοξενούσε την ετήσια τότε συνεδρίαση της Παγκόσμιας Τράπεζας και μιλούσαμε για το καθαρό νερό και για το καθαρό ουρανό για το περιβάλλον της Κίνας που ήταν πάρα πολύ υποβαθμισμένο λόγω της οικονομικής ανάπτυξης τότε. Και υπολογίσαμε ότι το, οικονομικό, μάλλον το οικολογικό το κόστος ε, της ρήπανσης στην Κίνα ήταν ε, μέχρι 8% του ΑΕΠ. Το συζητήσαμε λοιπόν με την κινέζικη ηγεσία. 8% ε, ήταν τότε η ρυθμή ανάπτυξης της οικονομίας αλλά και 8% έχαναν λόγω αυτού του γεγονότος. Και ε, αυτό το εύρημα συζητήθηκε επί εβδομάδες, εβδομάδες, εβδομάδες και τελικά το βάλαν σε μία υποσημείωση. Ότι α, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα λέει το κόστος είναι 8% του ΑΕΠ. Αλλά έδωσαν προσοχή και μπορώ να σας πω γιατί το έχω δει έκτοτε και έχω δει τεράστια αλλαγή στη συμπεριφορά του Σήμερα μας ξεπερνάνε στην παραγωγή ηλιακών ε, ε, συλλεκτών. Λοιπόν, για να μην πολύ λόγο. Θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες πολλές και το είπε και ο κύριος Κάσμεν και συνέπεια και διασύνδεση. Γίνονται αυτά. Το δικό μας πρόβλημα είναι ότι δεν γίνονται με την ταχύτητα που θα θέλαμε και εσείς ως βουλευτές είστε οι καλύτεροι μας φίλοι, διότι ε, κινείτε αυτά τα νήματα, κάνετε αυτές τις συζητήσεις και έχετε και την πολιτική ισχύ να επιταχύνετε αυτό που κάνουμε εμείς. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Νομίζω ότι ολοκληρώθηκε αυτό το τμήμα της ε, συνεδρίασής μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συζητητές μας ε, για την εξαίρετη ανταλλαγή απόψε που είχαμε. Σας ευχαριστούμε.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 Merci beaucoup, beaucoup. Merci. On Merci les jambes. Bye, Merci Bye. It's really not good to stand up. de se Nous allons continuer, surtout ne pas... Θα συνεχίσουμε, μην φεύγετε σας παρακαλώ, λέει η Πρόεδρος. Alors, ce qui... Si possible, rester dans la salle est encore mieux. Λοιπόν, το καλύτερο είναι να μείνετε στην αίθουσα, αλλά αν έχετε αποφασίσει να φύγετε, τουλάχιστον να φύγετε ησύχως. Θα κάνουμε τώρα παρουσίαση της ε, έρευνας την οποία έχει ζητήσει η Επιτροπή μας σχετικά με την εκτίμηση επιπτώσεων της διεκτησίας γης και της αρπαγής γης στην ανάπτυξη. Θα θυμάστε φαντάζομαι ότι η Επιτροπή μας είχε οργανώσει εδώ και ένα χρόνο τον Ιούνιο του 2010 μία ακρόαση για το θέμα αυτό και ο συνάδελφός μας ο κύριος Ντέβα ε, προετοίμασε από ε, αυτού του θέματος ε, ένα, μια έκθεση πρωτοβουλίας η οποία θα παρουσιαστεί και θα συζητηθεί σύντομα. Τώρα η, έκθεση είναι έτοιμη και θα συζητήσουμε λοιπόν το θέμα αυτό και τα αποτέλεσμα της έκθεσης με την κυρία Κριστίν Γκερστέτερ από το Ινστιτούτο Ecologic της Γερμανίας και τον κύριο Ζωάν Φιλίπ Πλατό από το Πανεπιστήμιο Notre Dame de la Paix. Είναι οι δύο που έχουν εργαστεί για το θέμα αυτό. Τους ευχαριστώ που είναι μαζί μας σήμερα για να μας παρουσιάσουν τα κεντρικά σημεία αυτής της έρευνας. Θα δώσω αμέσως τον λόγο στην κυρία Γκέρ Στέτερ, που θα είναι η πρώτη που θα μιλήσει. Well, good afternoon, ladies and gentlemen. Καλής, καλό σας απόγευμα και ευχαριστώ που μας καλέσατε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Επιτροπή σας για τη δυνατότητα που μας δώσατε να εγκύψουμε στο ενδιαφέρον αυτό θέμα που είναι και σημαντικό και επίκαιρο αλλά και περίπλοκο και τόσο περίπλοκο έχουμε καταλήξει, αυτό δείχνει ότι έχουμε καταλήξει να γράψουμε 30 σελίδες ενώ είχαμε ξεκινήσει από μια ιδέα να γράψουμε 10 μόνο σελίδες για τη μελέτη αυτή αλλά βέβαια τα πράγματα αυτά είναι σε βάση στοιχείων που συλλέγονται εδώ και 4 δεκαετίες. Τώρα, ο Ζαν Φιλίπ Πλατό είχε την καλοσύνη να αναθεωρήσει τη μελέτη μας. Είναι οικονομολόγος ειδικευμένος στην ανάπτυξη και έχει ασχοληθεί με τα θέματα της έγκυας ιδιοκτησίας. Εγώ θα παρουσιάσω τη μελέτη και ο συναδελφός μου, κύριος Πλατώ, θα συζητήσει μετά ε, μαζί σας. Θα παρουσιάσω πρώτα δύο βασικά αποτελέσματα της ε, μελέτης μας, ε, πρώτα από τα πιο αμφιλεγόμενα για τις επίσημα κατοχυρωμένα, τα επίσημα κατοχυρωμένα επίσημα κατοχυρωμένες ιδιοκτησίες, επίσης ποιες είναι οι επιδράσεις τους και οι αγορές και ούτω καθεξής ε, γηπέδων. Η σημασία της γης για την ανάπτυξη είναι γνωστή η πρόσβαση στην γη είναι σημαντικό εργαλείο για τη μείωση της φτώχειας. Ορισμένες μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι σε χώρες όπου είναι πιο δίκαιη η κατανομή της γης είναι και μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη, αν και οι αιτιώδεις συνάφειες για την ώρα δεν είναι σαφείς. Παρά τα θετικά αυτά στοιχεία του τι μπορεί να κάνει η γη δηλαδή για τη μείωση της φτώχειας. Πολλές αναπτυσσόμενες χώρες ε, πλήττονται από άνηση κατανομή. Πολλές μικρές εκμεταλλεύσεις έχουν πολύ μικρές ε, γης ενώ μεγάλα τμήματα γης είναι συγκεντρωμένα σε λίγα χέρια. Επίσης, στις αναπτυσσόμενες χώρες η πρόσβαση στη γη δεν είναι ε, αυτόματα ατομικό δικαίωμα, αλλά είναι σε τελείως διαφορετικές ε, σχέσεις. Υπάρχουν δηλαδή ε, άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται στη γη, δουλεύουν τη γη, αλλά με απλή ανοχή των κρατικών αρχών και ούτω καθεξής. Είπα ότι υπάρχει συνένεση σχετικά με την σημασία της γης για την ε, ανάπτυξη, αλλά δεν υπάρχει συνένεση σε ό,τι αφορά το πώς θα επιτευχθεί αυτό. Ένα άλλο ζήτημα είναι των δικαιωμάτων έγκαιας ιδιοκτησίας. Έχει προβληθεί το επιχείρημα και προτείνεται κυρίως από τον Ενάντο Ντεσότο, περουβιανό οικονομολόγο, που λέει ότι για να βγουν οι φτωχοί από τη φτώχεια πρέπει να τους δοθεί η ιδιοκτησία, η κυριότητα των ε, περιουσιακών στοιχείων, δηλαδή και ε, γη αλλά και σπίτια κλπ. Ο Ενάντο Τουσότο αναμένει από μια τέτοια εξέλιξη τρία πράγματα. Πρώτο, ότι οι τίτλοι ιδιοκτησίας θα αυξήσουν την επένδυση στη γη, άρα θα αυξηθούν οι δραστηριότητε. Αυτό θα γίνει διότι εάν οι άνθρωποι έχουν μια μακροπρόθεσμη προοπτική για την γη που του ανήκει, είναι πιθανότερο να επενδύσουν, ενώ αν γνωρίζουν ότι θα του πετάξουν έξω σε λίγα χρόνια, δεν θα το πράξουν. Πρώτο επιχείρημα αυτό. Δεύτερο επιχείρημα είναι ότι οι επίσημοι τίτλοι κυριότητα θα του επιτρέψουν και πρόσβαση σε δανειοδοτήσεις, χρησιμοποιώντας ως ασφάλεια υποθήκη δηλαδή τη γη τους, και θα αναπτυχθεί και σχετική αγορά. Δηλαδή οι τίτλοι ιδιοκτησία θα μπορούν να απολούνται και να αγοράζονται από αυτούς που θα δουλέψουν τη γη με αποτελεσματικότερο τρόπο. Τα αποτελέσματα αυτά έχει φανεί ότι λειτουργούν, ε, ότι ε, προκύπτουν δηλαδή σε ορισμένες χώρες ή υπό ορισμένες συνθήκες, αλλά έχει ασκηθεί και πολύ κριτική. Ο Ντεσότο και η Συναυτό έχουν επικριθεί επίσης σημαντικά γιατί υπάρχουν και μελέτες που δείχνουν ότι και αυτές οι κριτικές ισχύουν. Άρα η συνολική εικόνα είναι περίπλοκη και δεν υπάρχουν αυτονόητες συνταγές. Η διασύνδεση ανάμεσα στην ε, κατοχή τίτλων, τίτλων ιδιοκτησίας και την παραγωγικότητα δεν είναι αυτονόητη. Υπάρχουν και ενδείξει ότι ορισμένες φορές η τίτλοι διοκτησίας δεν είναι καν καλοί για του φτωχού, διότι του οδηγούν σε αυτά που λέγονται στα αγγλικά distressed sales, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες, για παράδειγμα λόγω φτωχή εισοδιά, θα πουλήσουν την γη του για να αγοράσουν τρόφιμα ή φάρμακα. Εν τέλει δεν θα έχουν λοιπόν στα χέρια τους ούτε την ε, γη, αλλά ούτε και χρήματα άρα θα, έχουν, ε, ε, θα βρίσκονται σε χειρότερη κατάσταση μακροπρόθεσμα. Τέλος, το κόστος για την κτήση τίτλων κυριότητας είναι σημαντικό. Υπάρχουν μελέτες οι οποίες υπολογίζουν ότι το κόστος για την κτήση τίτλων ιδιοκτησίας είναι μεγαλύτερο από τα προσδοκόμενα κέρδη και επομένως πολλοί οι οποίοι θα μπορούσαν να καταχωρήσουν τίτλους ιδιοκτησίας προτιμούν να μην το πράξουν. Υπάρχουν και θέματα εθνικού δικαίου που δεν μπορούν να αγνοούνται από τους ε, οπαδούς της ε, θεωρίας της, των, τίτλων, των τίτλων ιδιοκτησίας. Από την άλλη μεριά πολιτιστική λόγοι μπορούν να οδηγήσουν στη μη δυνατότητα πώληση της ε, γης, για παράδειγμα, όταν ε, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να επιτύχει να ζητήσει και να επιδιώξει την άδεια των μελών της οικογένειας του για να το πράξει. Το ίδιο ισχύει για το ότι ε, οι τίτλοι διοικησίας καταχωρίζονται συνήθως στο όνομα αρένων μελών της ε, οικογένειας και αυτό προκαλεί δυσχέρειες στην περίπτωση που ε, καλούνται οι γυναίκες να εκμεταλλευτούν την έγκαια ιδιοκτησία. Εν τέλει, κάτι που έχει γράψει ο Δεσότο πάλι στην ιστορία του κεφαλαίου που δεν αναφέρεται στην κατανομή των γεών αλλά στη σημασία της γης για τους στοχούς και που λέει για την άνηση κατανομή της, γε, της γης που είναι πολύ σημαντικό για τους αναδασμούς. Ολοκληρώνοντας το μέρος αυτό για την σημασία δηλαδή των τίτλων ιδιοκτησίας της γης δεν υπάρχει και καμία λύση ομοιόμορφη για όλους. Η τίτλη ιδιοκτησίας είναι μέρος της λύσης, αλλά δεν είναι η μοναδική λύση και θα πρέπει να συνοδεύονται και από λήψη άλλων μέτρων. Οποιοδήποτε, οποιαδήποτε ε, δραστηριότητα αναδασμού θα πρέπει να συνοδεύεται και από άλλα μέτρα που να επιτρέπουν την ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων, το λεγόμενο capacity building, επίσης τα, των δικαιωμάτων ε, για την άρτευση, τα νερά δηλαδή, και κυρίως για να μπουν στην εκμετάλλευση άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν, δεν έχουν δηλαδή κάνει, δεν έχουν αξιχεί τα δραστηριότητα αυτή στο παρελθόν. Υπάρχουν ωστόσο και ενδείξεις ακόμα ότι η ασφαλής πρόσβαση στην, στις είναι σημαντικότερη και από την ύπαρξη επίσημα καταχωρισμένων τίτλων ιδιοκτησίας. Αυτά για το πρώτο μέρος της μελέτης μας. Στο δεύτερο Μιλούμε για τις ε, μεγάλες κτίσεις γεών, την αρπαγή γεών δηλαδή, το land grabbing. Θα σας αναφέρω τα επιχειρήματα όσοι έχουν για την ώρα και μπορείτε να εξετάσετε και τη μελέτη για να δείτε τις λεπτομέρειες. Υπάρχει και κάποια συζήτηση που διεξάγεται σχετικά με τους κινδύνους και τις ευκαιρίες του λεγόμενου land grabbing για την ανάπτυξη. Η οι μη κρατικέ οργανώσεις ανησυχούν ε, από την εξέλιξη αυτή για την παραγωγή τροφίμων, διότι χρησιμοποιούνται γέες για την παραγωγή τροφίμων, τα τρόφιμα αυτά όμως εξάγονται σε άλλες χώρες, οι γέες αυτές που αποκτώνται ε, χρησιμοποιούνται για την παραγωγή φυτών για βιολογικά καύσιμα. Μέχρι τώρα, ωστόσο, η έρευνα δεν έχει γίνει σε βάθος και συχνά πάντως οι τίτλοι έγκες ιδιοκτησίας συνοδεύονται και από τους τίτλους ε, παροχής ε, υδάτων άρδευσης. Τέλος, και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ένα θέμα, το δικαίωμα στην τροφή. Το ερώτημα επίσης, και αυτό είναι το δεύτερο μέρος, πώς η πρόσβαση των τοπικών γεωργών ε, επηρεάζεται από μεγάλες αγοραπολισίες γεών. Οι άνθρωποι που ζουν από τη γη πιθανόν να μην είναι αυτοί που έχουν τους επίσημα καταχωρισμένους τίτλους. Εάν λοιπόν η κυβέρνηση εκχωρεί γέες που επίσημα είναι ιδιοκτήτης τους, δεν λαμβάνει υπόψη τα δικαιώματα αυτά τα οποία δεν είναι επίσημα καταχωρισμένα. Και οι τοπικοί γεωργοί μπορούν να χάσουν τις γέες τους και αυτό μάλιστα έχει διαπιστωθεί σε ορισμένες περιπτώσεις. Επίσης, αδύναμα νομοθετικά πλαίσια για τις ε, κτήσεις γεών, έλλειψη ε, παρακολούθησης και δημοσιοποίησης και με δυσκολία μάλιστα και για τους ε, ντόπιου, γεωργούς και άλλους, να έχουν πρόσβαση στις ε, απαραίτητες πληροφορίες. Και εν τέλει, ένα σημαντικό είναι η απώλεια της ρυθμιστικής ικανότητας των ε, χωρών υποδοχής για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Διότι συχνά εκχωρούν τις γέες με μακρόχρονες μισθώσεις και μιλούμε για 50 ή 100 χρόνια. Και αυτό είναι επιβλαβές για την ε, τοπική ανάπτυξη διότι η φιλοξενούσα χώρα δεν έχει τη δυνατότητα ή έχει πολύ περιορισμένη δυνατότητα ανατροπής της σύμβασης και κυρίως εφόσον η σύμβαση αυτή έχει ε, γίνει αντικείμενο πρόχειρης διαπραγμάτευσης και δεν προβλέπει σχετικές ρήτρες. Επίσης, κατά τη γνώμη ορισμένων, η Παγκόσμια Τράπεζα και ορισμένες ε, αναπτυσσόμενες χώρες μέλη, οι κυβερνήσεις τους δηλαδή, ε, θεωρούν θετικές τις αλλοδαπές επενδύσεις για τη δημιουργία απασχόλησης, για τη βελτίωση της υποδομής και της τεχνολογίας. Ορισμένες από αυτές τις ε, συμφωνίες αγοραπολισίας γεών περιλαμβάνουν και ρήτρες ότι ο αλλοδαπός επενδυτής θα πρέπει να κάνει επενδύσεις στην υποδομή ή στην δημιουργία απασχόλησης, αλλά το ρυθμιστικό πλαίσιο συνήθως είναι πάρα πολύ ασθενές και αυτό, όπου συμβαίνει αυτό, είναι πολύ απίθανο ε, τα αποτελέσματα αυτά πραγματικά να υλοποιηθούν. Για την ώρα πάντως δεν υπάρχουν ακλόνητα στοιχεία, οι πρώτες μελέτες οι οποίες ε, προχωρούν σε συστηματική, σε συστηματική εξέταση του τι συμβαίνει, τώρα συντάσσονται. Πολλές από τις συμφωνίες αυτές έχουν γίνει στα χαρτιά, αλλά η εφαρμογή τους δεν έχει ακόμη αρχίσει. Είναι λοιπόν πρόημο να πει κανείς οτιδήποτε για το τι θα γίνει. Νομίζω ότι τα πιο σημαντικά είναι αυτά για το λεγόμενο policy brief. Θα δώσω το λόγο στους υπόλοιπους προσκεκλημένους, αν θέλετε να μιλήσετε. Ο κύριος Πλατό. Do we answer to questions or maybe it is better? Okay, oh, donc d'abord. Μάλιστα. Αν θέλετε να συνοψίσω, να μιλήσετε και σε, στο μικρόφωνο. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Yes, Θα είμαι πάρα πολύ σύντομο στο παρόν γιατί το σημαντικότερο είναι να ακούσουμε τις δικές σας ερωτήσεις και να απαντήσουμε τα συγκεκριμένα θέματα που σας ενδιαφέρουν. Αυτό που είναι γνωστό ως αρπαγή γης, είναι κρίσιμο τώρα γιατί καλπάζει. Και όχι μόνο καλπάζει, αλλά και συγκεκριμένες περιοχές. Δεν είναι ευρέω διαδεδομένο παντού, είναι σε συγκεκριμένες περιοχές. Μέχρι τώρα έχει δοθεί ε, ε, μεγάλη προσοχή ε, ε η αγορά γης από κράτη, ιδιαίτερα σε αναπτυσσόμενες χώρες, οι Ινδοί γνωρίζουν πολύ καλά ότι συμβαίνει και στο εσωτερικό των ίδιων των χωρών αυτών. Και κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τις διασυνοριακές διεθνείς ε, περιπτώσεις αρπαγής γης. Αυτό ήταν το πρώτο ε, που ήθελα να σας πω. Το δεύτερο είναι το εξής. Αυτό τον καιρό γίνεται μια συζήτηση και ε, πραγματικά μας προξενεί εντύπωση ότι όλα αναφέρονται σε υποθετικό χρόνο, γιατί δεν έχουμε τα πραγματικά περιστατικά και στη βιβλιογραφία και στις συζητήσεις, όλα γίνονται σε υποθετικό λόγο. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει επί τόπου, γιατί μέχρι τώρα δεν έχουμε συστηματικές μελέτες που να ε, μετρούν μετά από κάποια χρόνια τον αντίκτυπο των επενδύσεων που γίνεται, γιατί χρειάζονται κάποια χρόνια ε, η απάντηση είναι ε, και τι να κάνουμε, να κάτσουμε και να περιμένουμε. Ε, και κάτι που είναι ανησυχητικό είναι ότι γνωρίζουμε τουλάχιστον ότι οι συμβάσεις ε, τις οποίες έχουμε δει είναι πάρα πολύ σύντομες και πάρα πολύ ασαφείς, αόριστες. Αυτό είναι το ανησυχητικό. Όταν βλέπετε αυτές τις συμφωνίες, οι διατάξεις που προστα προστατεύουν τους ντόπιου ε, χρήστες της γης είναι πάρα πολύ ασαφής και καθόλου λεπτομερής και γενικά ευσεβής πόθη. Αυτό θα πρέπει να μας ανησυχεί, διότι δεν ε, υπάρχει καμία δυνατότητα επιβολής του νόμου, κανενός είδους, ε, από κανένα φορέα, ούτε από το κράτος το ίδιο. Δηλαδή να υποχρεώσει κάποιον που έχει αναλάβει υποχρεώσει το διεθνή, τον ξένο επενδυτή, να τη στηρίσει κιόλας. Uh... Αυτό θα πρέπει να μας ε, κρούει ένα κόδωνα κινδύνου. Βεβαίω δεν χωράει καμία αμφιβολία, και γιατί να το κρύψουμε άλλωστε, ότι γίνεται πολύ μεγάλη ε, χρήση ε, μάλλον υπάρχει ε, η αρπαγή σε πόρους που υποχρησιμοποιούνται ή δεν τους εκμεταλλεύονται και υπάρχει ε, μεγάλη ε, σπατάλη ας πούμε ή χαμένο γιατί πρέπει να χρειαζόμαστε Κινέζους, Λίβιους ή κάποιους άλλους για να, να χρησιμοποιούν τη χώρα. Στη Βραζιλία γιατί ολόκληρα σε εκτάσεις παραμένουν ε, χέρσες και πρέπει να έρθουν οι Κινέζοι να τις καλλιεργήσουν. Γιατί ε, ε, ο οργανισμός του Νίγηρα στο Μάλι ας πούμε πρέπει να δραστηριοποιηθεί γιατί έχουμε εκατοντάδες και χιλιάδες εκτάρια ανεκμετάλλευτα χέρσα που δεν καλλιεργούνται και δεν αναπτύσσονται Why is it so? γιατί γίνονται όλα αυτά, γιατί συμβαίνουν γιατί πάει χαμένο τόσο νερό στον Ήγυρα που να είναι πρόβλημα για τον τοπικό πληθυσμό και τους αγρότες. Γιατί δεν απαντάει κανείς αυτό. Και όταν βλέπετε μια κυβέρνηση που πουλάει ή εκποιεί ή παραχωρεί τη γη για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, για πολλά χρόνια σε ξένες ε, ε, ξένους φορείς με πάρα πολύ ελαφρία συμβόλια αντί να παίρνει πρωτοβουλία και να εκμεταλλεύεται και να αξιοποιεί το ίδιο το κράτος ε, με άμεσες ξένες επενδύσεις. Για μένα είναι αυτό πρόβλημα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέχεται, γιατί υπάρχουν και Ευρωπαίοι επενδυτές εκεί. Βέβαια, θα πρέπει να ομολογήσω ότι δεν είναι η σημαντικότερη από, από πλευρά συμμετοχή. Είναι και άλλες οι χώρες που είναι ε, μη ευρωπαϊκές. Αυτά. Πάντως η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τώρα υποστηρίζει τη γεωργία ας πούμε, σε φτωχές χώρες της Αφρικής η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά θα πρέπει να ανησυχούν και να κοιτάνε τι γίνεται με τις καλλιεργήσιμες γέες και με κάποιο τρόπο να συζητούν ε, για τη χρήση γεών με την κυβέρνηση. Πώς θα γίνει αυτό να το συζητήσουμε μαζί σας. Αλλά είναι κάτι που δεν μπορούμε να το αποφεύγουμε πλέον. Ιδιαίτερα γιατί είναι λίγες οι χώρες αυτές που ενέχονται στην υπόθεση. Ευχαριστώ. Οι βουλευτές έχουν το λόγο. Η κυρία Κέλλερ πρώτη. Ευχαριστώ. Και για την παρουσίαση αυτή. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η μελέτη. και αυτό το θέμα της χρήσης γης. Είναι κάτι που έχουμε συζητήσει εδώ επανειλημμένα σε εκθέσεις μας και νομίζω ότι πολλοί ήταν υπέρ αυτής ε, της άποψης που λέει ότι όταν κάποιος κατέχει, ε, έχει αγοράσει τη γη, είναι αυτοκίνητρο για επενδύσεις, κρίμα που έφυγε ο κύριος Δέβα. Ε, διάβασα την έκθεση αυτή και τη μελέτη όπως και άλλοι. Είναι πολύ σημαντικό ε, να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία. Πολύ λογικά ακούγονται τα επιχειρήματα. από άλλες χώρες, ας πούμε, και άλλους πολιτισμούς και κουλτούρες και ανατροπίες, αλλά θα πρέπει να έχουμε και την ε, απόδειξη όλων αυτών που ακούμε κάποιοι να ισχυρίζονται γιατί μπορεί τα πράγματα μην είναι όπως φαίνονται. Αυτό ήταν το πιο ενδιαφέρον από την ε, μελέτη σας και θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Αλλά δεν είναι πάντα μηχανικός αυτοματισμός. Στο μέλλον θα το κοίταω έτσι πιο επικριτικά αυτό το επιχείρημα. Και για την υπόλοιπη μελέτη ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά ε, τους μηχανισμούς διεθνούς διακυβέρνησης. Ενδιαφέρον βρίσκω αυτό που λέγεται ότι επικρίνεται πολύ τις ε, αρχές που έχουμε που δεν είναι δεσμευτικές και λέτε θα πρέπει να ενισχυθούν παρόλα αυτά. Μα πώς, όταν οι συμφωνίες δεν είναι δεσμευτικές και είναι προαιρετικές και είναι θελοντικές και είναι ιδιαίτερα ανίσχυρες, ποια θα ήταν η διαφορετική λύση, πώς θα κάναμε ένα μηχανισμό πιο δεσμευτικό. Και εμεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πώ θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν ξέρω, όχι μόνο σε επίπεδο Ένωση, αλλά και σε επίπεδο κρατών μελών. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε που να είναι δεσμευτικό λοιπόν και να αφορά τουλάχιστον εταιρείε που αγοράζουν τη γη και να είναι κοινοτική ε, ιδιοκτησία ε, μερικώ ή ε, εξ ολοκλήρου. Ή τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε να μερικό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη είπατε ότι δεν γνωρίζουμε πολλά για τον αντίκτυπο. Γιατί ήθελα να ρωτήσω. Ξέρουμε πόσες θέσεις απασχόλησης ντόπιων γεωργών δημιουργήθηκαν. Φαντάζομαι δεν θα μπορέσετε να μας δώσετε απάντηση. Και κάτι άλλο που μας κάνει εντύπωση είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας. Γιατί ακούμε πάντα από τις κυβερνήσεις το κάνουμε γιατί θέλουμε να έχουμε την πράσινη επανάσταση, με την ε, πράσινη οικολογική, με την πιο πρόσφατη τεχνολογία. Και αυτό λειτουργεί. Γιατί όταν έρχεται κάποιος και αρπάζει τη γη ε, και μια εταιρεία αγοράζει ένα τεράστιο αγρόκτημα, φαίνει την τελευταία τεχνολογία, αλλά τη χρησιμοποιεί μόνο στο εσωτερικό του αγροκτήματος. Και οι διπλανές καλλιέργειες τι θα γίνουν, οι διπλανές εκμεταλλεύσεις που είναι και μικρής κλίμακας, γιατί μπαίνουν και ζητήματα οικονομικά εδώ. Υπάρχει δυνατότητα καν μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γκέρενς πρώτος. Merci, Madame la Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα βεβαίως να ευχαριστήσω τους ε, ομιλητές που αναφέρθηκαν σε αυτό το τόσο προφανώς επίκαιρο ζήτημα. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι το πολιτικό ζήτημα. Δηλαδή, τι μπορούμε να κάνουμε απέναντι σε αυτό το φαινόμενο. Πώς μπορούμε να απαντήσουμε ή να δώσουμε ένα προσχέδιο απάντησης. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να μάθω το εξής. Ποιοι είναι οι αγοραστές. Νομίζω ότι στην μεθοδολογία θα πρέπει να κάνουμε διαχωρισμό ανάμεσα στον θεσμικό αγοραστή και τον ιδιώτη αγοραστή. Υπάρχουν κράτη που εσκεμένα προσπαθούν να βάλουν το χέρι τους πάνω σε ε, γέες άλλων. Γιατί νομίζω ότι αν έχουμε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να θέσουμε ένα αμφιβόλο εταιρικέ σχέσεις που ενδεχομένως έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις χώρες αυτές. Για, θα πρέπει δηλαδή για τις αναπτυσσόμενες χώρες να αποτελέσει ένα, μια προϋπόθεση αιρεσιμότητας ε, αυτού του είδους η πρακτική, έτσι ώστε σιγά σιγά να βρεθεί μια λύση για το ζήτημα αυτό. Εάν πρόκειται για θεσμοθετημένη πολιτική κρατών, αυτό βεβαίως θα πρέπει να είναι πρόβλημα για μας. Και ποιες είναι οι πληροφορίες μας ε, ή τι μπορείτε να μας πείτε πάνω στο θέμα αυτό. Η δεύτερη κατηγορία είναι οι ιδιώτες αγοραστές. οι οποίοι κάνουν ό,τι θέλουν, κινούμενοι σε, ένα, κινούμενοι σε εδάφη ε, όπου έχουν απόλυτη ελευθερία, δεν είναι υπόλογοι σε κανέναν. Μπορούν να αγοράσουν λοιπόν γες. Και φαντάζομαι ότι αυτό συμβαίνει σε χώρες ε, με κακή διακυβέρνηση, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούσε να γίνει. Αναφέρομαι ας πούμε σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες μέχρι πρόσφατα ε, άσκησαν ε, μια συγκεκριμένη πολιτική ε, για να διατηρήσει την έγκαιη ιδιοκτησία στα χέρια των δικών της πολιτών. Ξέρω ότι η Γαλλία, ας πούμε, ήταν μία από αυτές τις χώρες, δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα σήμερα, πάντως ίσχυε μέχρι πρόσφατα. και νομίζω ότι μπορεί να αποτελέσει ε, βάση προς για χώρες ε, αναπτυσσόμενες κυρίως, οι οποίες επιθυμούν να κρατήσουν τις γέες τους. Δεν καταλαβαίνω βέβαια, δεν ξέρω πολύ καλά τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. ξέρω ότι θα πρέπει να σταματήσει, ξέρω ότι πρέπει να σταματήσει αυτή η αδικία. Αλλά πώς θα τη σταματήσουμε την αδικία αυτή, με ποιο τρόπο θα κινηθούμε. υπήρχε αρχικά ο κώδικας ε, αρχών που έπρεπε να, μια συμπεριφορά που έπρεπε να ακολουθήσουν όλοι ε, όμως ο κώδικας αυτός ε, που δεν έχει έτσι πολύ, πρόκειται για κώδικες που δεν έχουν ε, μεγάλη δυνατότητα παρέμβασης. Στα Ηνωμένα Έθνη υπάρχει ένας κώδικας συμπεριφοράς που δίνει βέβαια την υποχρέωση διαφάνειας και ρίχνει φως σε κάποιες λεπτομέρειες, αλλά δεν είναι αρκετό. Ε, παρόλο που ξέρουμε ότι ακολουθείται κατά το μάλλον ή ήτον, περισσότερο κατά το ήτον παρά κατά το μάλλον, από τις διάφορες ε, κοινωνίες. Πάντως θα πρέπει να κάνουμε κάτι που πραγματικά να έχει αντίκτυπο στην ε, καθημερινή ζωή. Εάν δεν είμαστε σε θέση να ε, υποβάλουμε απτές προτάσεις τελικά δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία βασίζεται πράγματι σε συγκεκριμένες αρχές ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν θα είναι αυτή που θα πρέπει να ξεκινήσει και να βρει λύση στο πρόγραμμα. Έχει πολύ μεγάλη ηθική ευθύνη η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αν δεν ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πιστεύω να περιμένετε να ξεκινήσει η Κίνα, ας πούμε. Από εδώ θα πρέπει να ξεκινήσει η λύση. Κυρίως όμως ε, θα πρέπει να ε, καταδειχθεί από κάθε δυνατή κατεύθυνση η βούληση να συνεχίσουμε να ασχολούμαστε με το θέμα αυτό. Και euh, νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Μέχρι τώρα ε, πολλοί κάνουν διάφορα πράγματα γιατί δεν υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική αντίδραση, αλλά εμείς έχουμε ένα πολύ απτό θεσμικό σύστημα ε, και πρέπει να σκύψουμε πάνω στο θέμα αυτό. Και η ΦΑΟ ε, κάνει μελέτες πάνω στο ζήτημα αυτό ε, και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι μεγάλος ο αντίκτυπος και μεγάλες οι επιπτώσεις στην ανάπτυξη και στο εμπόριο, στις εμπορικές σχέσεις και στις εργασιακές σχέσεις. Και ξαναλέω ότι εάν δεν πάρουμε εμείς την πρωτοβουλία, δεν θα βρεθεί κάποιος άλλος και εγώ θα κάνω μια ερώτηση. Με πιο συγκεκριμένο τρόπο. Τι κάνουμε με την ΑΕΤ, πού βρισκόμαστε με την ΑΕΤ. Είδαμε το πρόβλημα της ιδιοκτησίας της γης, το πρόβλημα ε, των γεών, το πρόβλημα μάλλον ε, του, ότι δεν μπορέσαμε, δεν μπορέσαμε να καθαρίσουν ε, κάποια κομμάτια γης ε, γιατί οι ιδιοκτήτες ζούσαν στο εξωτερικό, ανήκαν λοιπόν ε, ανήκαν σε μέλη της διασποράς. Επίσης υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι εκμεταλλεύονταν τη γη πριν την καταστροφή και είδαν να χάνεται από τα χέρια τους η γη αυτή, αντιμετωπίσαμε πάρα πολλά προβλήματα στην IT. Τι κάνουμε λοιπόν. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Λιούινγκ και μετά θα απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη που ήμουν αργοπορημένη και δεν άκουσα ε, εξ ολοκλήρου τις παρεμβάσεις. Αυτή η αρπαγή γης είναι κάτι που με απασχολεί πάρα πολύ. Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τις αλλιευτικές συμφωνίες, συμφωνίες αλλιείας λοιπόν που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με πολλές ε, τρίτες χώρες και νομίζω και εκεί μπορεί να εφαρμοστεί η αρχή ε, μάλλον και εκεί βρίσκουμε αντίστοιχα προβλήματα. Δεν έχουμε αρπαγή γης, έχουμε αρπαγή υδάτων. Και νομίζω ότι θα πρέπει να συνδυαστούν τα δύο αυτά στοιχεία, αρπαγή γης και αρπαγή υδάτων. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ περίπλοκο ζήτημα. Όλοι λένε, εάν ε, δεν κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνίες αλληλείας ε, με άλλες χώρες, ε, είτε είναι η Γουινέα, είτε άλλες χώρες, τότε δεν θα έχουμε καμία δυνατότητα ελέγχου ε, ή δεν θα έχουμε επιστημονικές ε, εκτιμήσεις ε, για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η αλία και επομένως επαπειλείται η ασφάλεια της διατροφικής αλυσίδας. Έμαθα σήμερα για την, ναι, για την Κίνα ότι πρόσφατα έκανε μια συμφωνία εκείνη με την Μαυριτανία, συμφωνία διάρκειας 25 χρόνων, για πρόσβαση αναέτος σε 100.000 τόνους ε, αλλιεύματος. Βεβαίως λένε ότι θα χτίσουν ε, και κέντρα διαλογής ε, και we're talking about a, common resource. Και μεταποίησης ότι θα είναι δημόσιες, ε, δημόσιες αυτές οι ε, βιοτεχνίες και επομένως θα ανήκουν στην τωρινή και στη μελλοντική γενιά των Μαυριτανών. Το ζήτημα εδώ είναι να μπορέσει το Κοινοβούλιο να προκαλέσει συζήτηση έτσι ώστε όλα αυτά τα ζητήματα να υπόκεινται ε, στον ε, κοινοβουλευτικό έλεγχο, να υπάρχει διαφάνεια. Ε, ε, μου έρχεται στο μυαλό η πρωτοβουλία διαφάνειας των εξορρυκτικών διεργασιών και δραστηριοτήτων. Και όλα αυτά τα λέω γιατί θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Η διαφάνεια θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ καλή και για την περίπτωση των συμφωνιών αλληλείας για την αρπαγή υδάτων. Πιστεύετε ότι θα ήταν καλό και για την περίπτωση αρπαγής ε, ε γης. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούσε κάπως η κοινωνία των πολιτών να ασκεί κάποιον έλεγχο. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω πρώτα το λόγο τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον κύριο Σόμελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με μεγάλο ενδιαφέρον διαβάσαμε τη μελέτη αυτή που δείχνει πόσο περίπλοκο είναι το πρόβλημα. Πρέπει να σας πω ότι ήταν άριστη η μελέτη στην εκπόνησή της αλλά δεν βλέπω τίποτα για την κτηνοτροφία, την εκτατική τους βασκούς δηλαδή και τις γυναίκες. Ε, κατά τα άλλα συμφωνώ και συμμερίζομαι 100% με τα όσα λέτε. Ε, είναι περίπλοκο το πρόβλημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έχει συζητήσει από το 2002 με τα κράτη-μέλη. Εκπονήσαμε και έναν οδηγό για το πώς θα έχει η χρήση το 2004 και από το 2009 και μετά ε, επανεκκινήσαμε αυτή την προσπάθεια με τα κράτη-μέλη. Συνεργαζόμαστε πάρα πολύ και με το ΦΑΟ ε, για τον εθελοντικό οδηγό για τη χρήση των γεών. Δεν είναι εύκολο. Έχουμε από τη μια τα προβλήματα των επενδύσεων που είναι και ιδιωτικές και οι μη ιδιωτικές επενδύσεις και επίσης και το θέμα της ιδιοκτησίας της γης. Ε, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για σας ε, στη μελέτη σας είναι το συμπέρασμά σας. Το σημαντικότερο είναι η ε, εξασφάλιση της πρόσβασης εδώ εργαζόμαστε πάρα πολύ ε, για θέματα ιδιοκτησίας, κυριότητας γης, αλλά υπάρχουν στην Αφρική και αλλού ε, ζητήματα νοοτροπίας κουλτούρας, έτσι, και θα πρέπει να τα δούμε πάρα πολύ προσεκτικά. Πέρυσι ε, αρχίσαμε ένα πρόγραμμα σε συνεργασία, ένα έργο έτσι με την Αφρικανική Ένωση, για να αναπτύξουμε εθνικές πολιτικές υπέρ των γεών. Διότι συμφωνούμε με τη δική σας διαπίστωση ότι εάν δεν συμμετέχουν και οι χώρες που είναι συνομιλητές και εταίροι μας, θα υπάρχει μεγάλη δυσκολία να προχωρήσουμε. Επίσης, η κοινωνία των πολιτών και οι κοινότητες παραγωγών, οι οργανώσεις παραγωγών πρέπει να συμμετέχουν. Σε αυτούς τους δύο πυλώνες εργαζόμαστε. Διαβάζω λοιπόν τη μελέτη και τις συστάσεις και διαισθάνομαι ότι ζητάτε να επιταχύνουμε λίγο τη λύση του προβλήματος. Το πρόβλημα είναι πολύ πιο περίπλοκο όμως. Αν κοιτάξετε την ευρωπαϊκή μας ιστορία, θυμάστε το θέμα των enclosures στην Αγγλία και κάποιος από τους ε, ιδρυτές της κοινή γεωργικής πολιτικής είχε πει «οι γέες να χαρακτηριστούν δημόσιο αγαθό και οι αρρώσιμες και οι μη αρρώσιμες. Ε, λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι είναι ιστορία μακρά και δεν είναι εύκολο να λυθεί το θέμα ε, γρήγορα. Η Ευρώπη ε, ήταν η πρώτη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρωτοστάτησε σε αυτή την προσπάθεια. Απλώς πρέπει να σας πω ότι οι λύσεις δεν είναι άμεσες, θα χρειαστούν πολλές συζητήσεις, να καταλάβουμε πάρα πολύ τι θέλουν οι συνομιλητές μας, οι χώρες και κυρίως οι πληθυσμοί τους. Χρειάζεται πολύ μεγάλη ενημέρωση. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξαναδώσω το λόγο με τη σειρά που θέλετε. Δεν ξέρω ποιος θέλει από τους δύο να αρχίσει. Thanks for the Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις και για τα σχόλια. Που έδειξαν άλλωστε πόσο ευρύ και περίπλοκο είναι το θέμα. Θα προσπαθήσω να απαντήσω. Η πρώτη ερώτηση για τους δεσμευτικούς ή μη μηχανισμούς. Στη μελέτη μας λέμε κάτι ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν μη δεσμευτικέ κατευθυντήρε γραμμέ, αλλά υπάρχουν τώρα και των δύο ειδών για τις ε, μεγάλες κτήσεις υγειών. Υπάρχουν investment guidelines και voluntary guidelines. Αυτές οι δύο διαδικασίε, εξετάζοντα οι δύο αυτές τις και τα έγγραφα που ε, παρήχθησαν και βρήκαμε ότι οι ε, ε, εθελοντικές κατευθυνές του ΦΑΟ συμβαδίζουν περισσότερο με τα δικά μας ευρήματα. Σε ό,τι αφορά ποιοι δεσμευτικοί μηχανισμοί μπορούν να προβλεφθούν, ένα από τα συμπεράσματα που, της μελέτης που δεν πρόλαβα να σας παρουσιάσω είναι για, το βιολογικό για τα βιολογικά καύσιμα και για τα κριτήρια αηφορίας που είναι ένας από τους παράγοντες που οδηγεί στις, ε, σε, μια έντονη τάση κτήσης μεγάλων ε, γεών. Είναι λοιπόν μια επιλογή όπου θα μπορούσατε να βάλετε κάτι ε, σημαντικό και δεσμευτικό ως στοιχείο στην υφιστάμενη νομοθεσία. Η άλλη επιλογή ε, για να στοχευτούν ιδίω Ευρωπαίοι επενδυτές ή μάλλον ευρωπαϊκές επενδύσεις είναι η ικανότητα λογοδοσίας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων για παραβιάση ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Αλοδαπή στο διεθνές επίπεδο θα ήταν επιθυμητό να υπάρχει ένα δεσμευτικό πλαίσιο. Από την άλλη μεριά με πολλές απόπειρες να γίνει διαχείριση των επενδύσεων στο διεθνές επίπεδο τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά δεν ήταν δεσμευτικές ε, συμφωνίες, εκτός από διμερείς μόνο, ή περιφερειακού χαρακτήρα, αλλά που είχαν μάλλον χαρακτήρα προστασίας των επενδυτών και λιγότερο προστασίας των δικαιωμάτων των ντόπιων πληθυσμών και του περιβάλλοντος τους. Η ιδέα λοιπόν να είναι δεσμευτικές οι κατευθυντήριες γραμμές για τις εκτίσεις γεών στο διεθνές επίπεδο δεν θα είναι μάλλον πολύ εφαρμόσιμη, αλλά για αυτά που είπα για τα βιολογικά καύσιμα, για τα κριτήρια βιωσιμότητας, για να είναι υπόλογες οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για το, κάνουν, για το τι κάνουν στην Ολοδαπή. Αυτά είναι πράγματα τα οποία γίνονται μονομερώς. Τι γνωρίζουμε τώρα για τις, ε, για τις ε, επιπτώσεις επιτόπου της αρπαγής γης. Η μελέτη του 2009 της Παγκόσμιας Τράπεζας διαπίστωσε ότι μόνο το 1 πέμπτο των συμβάσεων που είχαν ολοκληρωθεί στα χαρτιά είχαν αρχίσει να υλοποιούνται. Και για το λόγο αυτό, ένας από τους λόγους μάλλον, ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν γνωρίζουμε τόσα πολλά πράγματα είναι και η έλλειψη δεδομένων, την οποία ανέφερα και πριν. Υπάρχουν ωστόσο ορισμένε συμφωνίες οι οποίες περιλαμβάνουν ρήτρε σχετικά με τις δεσμεύσεις της, ε, των τοπικών κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων σε ορισμένες από τις συμφωνίες, αν και όχι σε όλες βέβαια, υπάρχει κάποιο σημείο αφετηρίας γι' αυτό. Σε ό,τι αφορά τις μεταφορές τεχνολογιών, αναμένεται να γίνει μεταφορά τεχνολογίας από τους ενδιαφερομένους, για παράδειγμα μοντέλων όπου η τοπική γεωργοί θα προσληφθούν από τους επενδυτές για να ε, παράγουν επιτόπου και να πολλούν τα προϊόντα τους στον επενδυτή και μέσα στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσε να τους ε, δοθεί τεχνολογία ή να χρησιμοποιήσουν άλλες τεχνολογίες από αυτές που χρησιμοποιούν συνήθως, άρα και αυτό θα ήταν μια μεταφορά τεχνολογίας. Αυτά θα μπορούσαν να συμβαίνουν, δεν είμαστε, να συμβούν, δεν είμαστε όμως βέβαιοι ότι θα συμβούν όντω. Υπήρχε και μια άλλη ερώτηση σχετικά με το εάν γνωρίζουμε ποιος προχωρεί σε αγορές γεών. Η ταυτότητα των αγοραστών γεών είναι γνωστή στο γενικό επίπεδο. Υπάρχουν ορισμένε μελέτες που προσπαθούν να συστηματοποιήσουν την γνώση για, στη βάση των υφιστάμενων συμφωνιών. Έχουν εντοπίσει τέσσερις βασικές ομάδες επενδυτών, εθνικές δηλαδή κυβερνήσεις, όμως αυτή είναι η σπανιότερη περίπτωση μετά τα ε, ταμεία δημόσιου χαρακτήρα, κυρίως των χωρών του Περσικού κόλπου, επίσης ιδιωτικές επιχειρήσεις, αλλά και κρατικού χαρακτήρα, δημόσιου χαρακτήρα επιχειρήσεις. Αυτές είναι οι τέσσερις βασικές ομάδες. Στη μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας, αλλά και σε άλλες μελέτες που έχουν γίνει στο ποσοτικό επίπεδο, διαπιστώνουν ότι περισσότερο είναι, οι περισσότεροι μάλλον είναι οι ιδιωτικοί επενδυτές από τους ε, δημόσιους. για το ρόλο των Ηνωμένων Εθνών. Ε, θα πει ίσως κάτι ο Φιλίππη γι' αυτό. Για την ΑΕΤ δεν είμαι σε θέση να σχολιάσω γιατί δεν γνωρίζω την κατάσταση στη χώρα αυτή. Για την αλληλεία ήταν ενδιαφέρον το ερώτημα. Νομίζω ότι είπα ότι η δημοσιότητα, η έλλειψή της είναι ε, σημαντικό χαρακτηριστικό Υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες αναπτύσσονται τώρα και όλες αναφέρονται στην ανάγκη δημοσιότητας και στην ενημέρωση των τοπικών πληθυσμών για τις ε, μεγάλες αυτές συμβάσεις κτήσης γεών. Εν τέλει, σχετικά με τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, νομίζω αναφερθήκατε σε ορισμένα από τα έγγραφα πολιτικής Εμένα με έχουν εντυπωσιάσει οι κατευθυντήριες γραμμές πολιτική, οι Land Policy Guidelines, που είναι μακροσκελές έγγραφο, αλλά δεν δίνουν συμβουλές του είδους ε, πρώτο βήμα, δεύτερο, τρίτο κτλ. Είναι πολύ ε, συνολική, είναι μάλλον ε, περιεκτική η προσέγγιση τους με τα διάφορα, με διάφορες πτυχές, αλλά δεν είναι ένα έγγραφο το οποίο να είναι και τόσο πολύ ε, γνωστό δημόσια. Έχουμε συνεργαστεί με τους ανθρώπους που εργάζονται στην ομάδα εργασίας για τις κτίσεις γεών. Πάντως, καταλήγω στο ότι, στην εντύπωση ότι ως όντας εκτός, ότι δεν είναι ένα έγγραφο το οποίο έχει διαδοθεί ευρέως. Και νομίζω ότι είναι καλό έγγραφο και θα μπορούσε να ε, διαδοθεί περισσότερο. Κύριος Πλατώ, ε, well informed and ε, in fact difficult question. σας ευχαριστώ πολύ, πολύ εμπεριστατωμένη και ενημερίστε. Ε, η γνώση σας είναι πολύ εμπεριστατωμένη και οι ερωτήσεις καθόλου εύκολες. Επιτρέψτε μου να απαντήσω. Ας επανέλθω σε αυτό το θέμα της κτήσης. Τι γνωρίζουμε σήμερα ότι σε πολλές φτωχές χώρες, ιδιαίτερα στην Αφρική, την υποσαχάρη Αφρική, ο κόσμος έχει άτυπα δικαιώματα, τίτλους, ιδιοκτησίας δεν έχουν. Δεν έχουν τίποτα γραπτό που να αποδεικνύει την ιδιοκτησία και το γνωρίζουμε αυτό και είναι πολύ δύσκολο να πούμε ότι εκείνοι που έχουν τίτλους ιδιοκτησίας έχουν πλεονεκτήματα έναντι αυτών που δεν έχουν. Στη Μαδαγασκάρη ε, ο Χάναν ε, Τζακόμπι τη Παγκόσμια Τράπεζα, έδειξε ότι ε, εκεί που έχουν γίνει έγκαιε βελτιώσει και αρδευτικά έργα και μεγάλες επενδύσεις, εκεί που έχουν τίτλους ιδιοκτησίας υπήρχαν όμως και ε, μικρά χωράφια ή κόπεδα χωρίς τίτλους. Αλλά δεν υπήρχε καμία διαφορά στη Μαδαγασκάρη πάντα. Ε, άλλες μελέτες και μεταξύ αυτών η κοπεδα χωρις τιτλους αλλα δεν υπηρχε καμια διαφορα στη μαδαγασκαρη παντα ε αλλες μελετες και μεταξυ αυτων οι δικοι μου έχουν δείξει ότι δεν είναι μεγάλη δυσκολία, δεν είναι πρόβλημα η έλλειψη τίτλων και για τη μεταβίβαση στα παιδιά τους κτλ. Έχουμε ε, δει και τέτοια ζητήματα όχι μόνο σε αγροτικές γεές αλλά και σε περιαστικές περιοχές. Και αυτό δεν είναι πρόβλημα. Πρόσφατα μελέτες στη Λατινική Αμερική ε, έδειξε ότι αν δώσετε σε άκληρους ε, αγρότες που, που λαμβάνουν τη γη τίτλους και τα παιδιά τους έχουν κληρονομήσει και τα σπίτια και τη γη, θα διαπιστώσετε ότι οι τίτλοι είναι σε λάθος όνομα. Και τι σημαίνει αυτό, ότι η επόμενη γενεά δεν ζήτησε να διορθωθούν ε, ε, τα ονόματα στους τίτλους ιδιοκτησίας στο ε, υποθικό φυλάκιο. Και η ερώτηση γιατί δεν γίνεται αυτό, η απάντηση είναι ε, γιατί είναι ακριβό. Δεν έχουν χρήματα να αλλάξουν το όνομα στους τίτλους. Λοιπόν, το σύστημα είναι έτσι κάπως άτυπο. Όπου δεν ξέρει ε, κανείς, αλλά οι ντόπιοι ξέρουν ποιανού γη, ε, σε ποιον ανήκει η γη. Εντάξει, για την ασφάλεια λέτε, για την πρόσβαση. Αυτό δεν ε, είναι εις βάρος του συστήματος. Εκτός αν είναι τόσο ακριβή η γη, ώστε να προσελκύει ξένους επενδυτές και τις επιβουλές του κράτους και τις ορέξεις. Αυτή είναι η κατάσταση. Και όχι επειδή ξαφνικά ανακάλυψε κάποιος ότι δεν έχουμε ε, ενέργεια ή καύσιμα ή ε, τρόφιμα. Ξαφνικά ορισμένε χώρες, άλλες κρατικές εταιρείες ε, ή υποτιθέμενες δημόσιες εταιρείες, αρχίζουν με κατανοητό τρόπο να εξασφαλίζουν τις προμήθειες τους και τα κράτη διαπιστώνουν ότι αυτές οι γέες που ήταν ε, εντάξει χωράφια των γεωργών για να επιβιώνουν ξαφνικά είναι μια ευκαιρία για το κράτος να αποκομίσει κέρδη. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι είναι πολύ μεγάλος πειρασμός για το κράτος να απαλωτριώσει κατά κάποιο τρόπο τις γέες αυτές και είναι εύκολο να απαλωτριωθούν διότι κανονικά ε, ο ε, ιδιοκτήτης, ο κύριος της γης, σύμφωνα με τον νόμο, και της γεωργικής γης είναι το κράτος και όχι η γεωργή. Γι' αυτό οι γεωργοί και οι αγρότες είναι ανυπεράσπιστοι. Και εκεί είναι το πρόβλημα. Και εκεί μπαίνουν κάπου οι διεθνείς οργανισμοί και η αναπτυξιακή βοήθεια. Εκεί θα πρέπει να ενταχθούν για να παίξουν κάποιο ρόλο. Αλλιώς η κατάσταση είναι πάρα πολύ αρνητική. Ένα δεύτερο που θέλω να πω. Το μοντέλο που ανέπτυξαν οι Κινέζοι στη Βραζιλία και σε κάποιες χώρες της Αφρικής δεν είναι κακό οι συμβάσεις. Εντάξει, είναι πολύ ωραία σύμβαση. Εσύ θες να εξασφαλίσεις κάποιες ε, προμήθειες, από την άλλη μεριά υπάρχουν οι αγρότες που δεν έχουν ούτε μέσα, ούτε τεχνολογία, ούτε τίποτα και πας και λες ότι κοίτα, πούλα μου το δικαίωμά σου να διαθέτω τη σοδιά και θα σε βοηθήσω να έχεις πρόσβαση στην τεχνολογία, σε σε δάνεια κλπ. Και γνωρίζουμε ότι αυτές είναι οι βασικές ε, δυσκολίες και περιορισμοί και στην Αφρική και σε απομακρυσμένες περιοχές της Λατινικής Αμερικής, ας πούμε στα υψίπεδα του Περού, όπου οι πολύ φτωχοί αγρότες δεν έχουν καμία πρόσβαση ούτε σε δάνεια, ούτε σε τεχνολογία. Είναι πολύ ακαθόδες το θέμα. Λοιπόν, ε, ε, έτσι, καταρχήν είναι καλές οι συμβάσεις τα συμβόλαια. Το πρόβλημα ποιος είναι, ότι το συμβόλαιο είναι καλό ε, στο βαθμό που έχουν τη δυνατότητα εξόδου καταγγελία οι αγρότε. Δηλαδή αν δεν τους αρέσει να, να το καταγγείλουν και να πάνε αλλού. Ε, εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Αν όμω έχουν το δικαίωμα, μάλλον ε, αν καταντήσουν να είναι μονοπόλιο που δεν μπορούν να βγουν γιατί το κράτος έχει νοικιάσει αυτή τη γη για 99 χρόνια, ε, υπάρχει μια παροχή και το ξέρουμε αυτό γιατί ε, περί ε, αυτής της περίοδου πρόκειται, από 49 μέχρι 99 έτη. Είναι πολλά χρόνια. Ε, δυο γενιές δεσμεύονται, ας πούμε, από αυτά τα συμβόλαια. Γιατί αυτό πια είναι επικίνδυνο, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα εξόδου. Και εκεί χρειάζεται παρακολούθηση και χρειάζεται και παρακολούθηση με μητρό, ο κόσμος να ε, παρακολουθεί τι γίνεται, να καταγράφει κάποια δυσφορία και να διορθώνει τα κακό κείμενα. Ελπίζω να απάντησα στην ερώτηση που έγινε προηγουμένως. Είπατε ότι ε, οι αγρότες θα πρέπει να διατηρούν ε, το μέσο παραγωγής τους και τη γη τους ναι, στα χέρια τους. Αλλά αυτό είναι το πρόβλημα. Τι σημαίνει τι γη είναι αυτή, υποβαθμισμένη. Πηγαίνετε στο Μαλί. Γιατί ο κόσμος πεινάει και πεθαίνει. Γιατί είναι πάρα πολύ υποβαθμισμένη η γη. Εάν θέλουν να τη διατηρήσουν, ωραία, ναι, να τη διατηρήσουν, αλλά να έχουν και ένα μέλλον γιατί είναι υποβαθμισμένη η γη τους, κατεστραμμένη και χρειάζεται να ε, ξανάρθει η γονιμότητα. Έρχονται οι Κινέζοι και σου λένε θα το κάνω εγώ, η κυβέρνησή τους δεν το κάνει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι ψελίζει, αλλά δεν φτάνει και αυτό. Ε, γιατί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χρησιμοποιεί αυτή τη δυνατότητα που έχει, πίεση τεράστια, για να κάνει αισθητή την παρουσία της, να πάει στην κυβέρνηση του Μαλή και να πει ότι ξέρουμε ότι αυτό το σύστημα δεν λειτουργεί σωστά, Και μάλιστα έχουμε βάλει και ένα σύστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταβλητό, εξαρτάται η εκταμείευση από το αποτέλεσμα και κρίνεται εκ του αποτελέσματο ε, που έχει επιτευχθεί ως τώρα η χώρα. Γιατί δεν το κάνετε, να πούμε ότι σα προσφέρουμε βοήθεια για να ενισχύσουμε τους μικροκαλλιεργητέ, αλλά με την προϋπόθεση ότι θα δημοσιεύσετε όλες τις συμφωνίες που κάνετε σε εκτάσεις, εντάξει με κάποιο μέγεθος έτσι, με ξένες εταιρείε και όπου υπάρχουν βάσιμοι φόβοι ε, ότι ε, θα είναι δυσμενήσεις οι βάσεις για τους αγρότες. Χρειάζεται κάποια πειθαρχία, κάποιες στρατηγικές για τους δωρητές και αυτό τον καιρό το συζητούν οι κοινότητες των δωρητών και για τη γεωργία. Εγώ δεν γνωρίζω πάρα πολλά πράγματα, αλλά εξ όσων μπορώ να κρίνω, Υπάρχουν κάποιες γιές που χαρακτηρίζονται προεδρικές γιατί είναι κρατικές και επειδή ο πρόεδρος της χώρας ε, αντιπροσωπεύει το κράτος θεωρούνται ότι είναι δικά του αυτά τα κτήματα. Ναι, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ εύθραστο και προσφέρεται για πολύ μεγάλη αυθαιρεσία από πλευράς του κράτους. Όχι. Μόλις αρχίζει λοιπόν να ενδιαφέρεται το κράτος για τη γη, για άλλη χρήση από καλλιέργεια, όσο δεν το ενδιαφέρει το αφήνει στον αγρότη. Αλλά θα πρέπει να προστατεύεται ο κόσμος. Και κάποιοι από την Παγκόσμια Τράπεζα στην αρχή διαφώνησαν μαζί μου. Ε, σε σχέση με τους επίσημους τίτλους και που έλεγα ότι δεν είναι τόσο σημαντικοί, τώρα έρχονται να συμφωνήσουν ότι χρειάζονται για να προστατεύονται οι ε, πολίτες από το ίδιο τους το κράτος. Ο Ερνάντο Ντεσότα, ας πούμε, το έχει καταλάβει πλέον ότι αυτό χρησιμοποιείται, οι τίτλοι χρειάζονται για να προστατεύονται οι αγρότες από τον ίδιο του τη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε θέση προνομιούχα και μπορεί να δράσει πάνω σε αυτό. Το θέμα για το ερώτημα είναι αν το πράττει. Και η σύγκριση με την αρπαγή της θάλασσας, των υδάτων και στην αλία είναι πολύ καλή. Η Βραζιλία τι έκανε. Ε, από ένα μέγεθος και πάνω δεν εμπόδισε κανένα να αγοράζει τη γη. Ε, ε, τώρα με τους Κινέζους την νοικιάζουν μόνο, δεν την πολλούν. Πλέον δεν, δεν μπορεί κανείς να αγοράσει κτήματα στη Βραζιλία, μόνο το νοικιάζει. Αλλά η Βραζιλία δεν είναι ούτε η Σιέρα Λεόνε ούτε το Μάλι. Άρα εμείς ως Ευρωπαίοι εδώ θα πρέπει να κάνουμε κάτι γιατί έχουμε ιδιαίτερη ευθύνη. Νομίζω ότι μπορώ να σταματήσω εδώ. Eh Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Σε ένα λεπτάκι θα συνεχίσουμε με την ημερήσια διάταξη. Voilà, Χωρίς ε, να χάσουμε καθόλου χρόνο, θα περάσουμε στο επόμενο θέμα που αφορά τη μελλοντική χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2014 μέχρι το 2020. Πέρσι το Κοινοβούλιο δημιούργησε μια ειδική επιτροπή η οποία ανέλαβε την εκπόνηση θέσεως του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εν ώψη των διαθεσμικών διαπραγματεύσεων. Το προηγούμενο μήνα η Επιτροπή αυτή, η ΣΟΥΡΕ, ψήφισε την τελική της έκθεση, η οποία εγκρίθηκε στην Ολομέλεια πριν από δύο εβδομάδες. Δύο μέλη της Επιτροπής μας συμμετείχαν στις εργασίες της ΣΟΥΡΕ. Οι συνάδελφοι Μπέρμανς, που δυστυχώς δεν είναι εδώ, και ο συνάδελφος Γκέρνς, που βεβαίως είναι εδώ. Η ΔΕΒ είχε επίσης ε, στείλει μια γνωμοδότηση στην Επιτροπή ΣΟΥΡΕ, η οποία όμω δεν έλαβε υπόψη τι προτάσεις τη επιτροπή ανάπτυξη. Παρ' όλα αυτά, η έκθεση της ΣΟΥΡΕ περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο για την ανάπτυξη. Λαμβάνοντας υπόψη την ε, σημασία των διαπραγματεύσεων για το επόμενο χρηματοδοτικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόταση θα δημοσιευθεί τη 20 Ιουνίου 2011, αποφασίσαμε να οργανώσουμε νέα ανταλλαγή απόψεων σήμερα όσον αφορά τα αποτελέσματα της εργασίας της ΣΟΥΡΕ. Χαίρομαι που η συγητής Επιτροπής ΣΟΥΡΕ, όπως ε, ο κύριος ε, δηλαδή Σαλβαδόρ Καρδίγκα και η κύριοι Φέρμ και Καρίσα Ντάλ θα είναι μαζί μας ε, και έχουν αποδεχθεί την πρόσκληση να βρίσκονται μαζί μας. Θα τους δώσω αμέσως το λόγο, έτσι ώστε να ακούσουμε την εκτίμηση που θα μας δώσουν για το τελικό αποτέλεσμα της ΣΟΥΡΕ, κυρίως τα θέματα που ε, αναφέρονται σε θέματα ανάπτυξης. Muchas gracias, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. δεν πειράζει για το επίθετο. Εδώ στο Κοινοβούλιο όλοι περίεργα ονόματα έχουμε ε, και δυσκολίες στην προφορά. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Ανάπτυξης για την πρόσκληση που μας απίφθηνε σας εξηγήσουμε λίγο πώς πήγαν οι εργασίες της Επιτροπής ΣΟΥΡΕ και να κάνουμε μια μικρή ανταλλαγή απόψεων. Υποθέτω ότι και η Επιτροπή σας, όπως οι περισσότερες επιτροπές και οι περισσότερες πολιτικές ομάδες, δεν είμαστε 100% ικανοποιημένοι από την έκθεση. Αλλά είναι προφανές ότι ένας από τους στόχους ήταν να μπορέσουμε να κάνουμε μια έκθεση που να εγκριθεί κατά πλειοψηφία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι διάφορες επιτροπές της νομοδοτήση τους αλλά και οι πολιτικές ομάδες αναγκαστήκαμε να εγκαταλείψουμε κάποια αιτήματα για να καταλήξουμε σε ένα γενικό συμβιβασμό και σε μια γενική συμφωνία. Βεβαίω η Επιτροπή Σούρε δέχτηκε και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής σας, της Επιτροπής Ανάπτυξης. Και φαντάζομαι ότι δεν θα είδατε όλα σας τα αιτήματα να γίνονται δεκτά. Αλλά θα ήθελα να σας πω ότι η έκθεσή μας ήταν αρκετά γενικόλογη. Και ο στόχος μας να δούμε λίγο και να καθορίσουμε τις στατικές γραμμές προς τα που θέλαμε να κατευθύνεται η έκθεση των δημοσιονομικών προοπτικών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν θέλαμε να μπούμε ούτε σε λεπτομέρειες και ούτε ε, ασχοληθήκαμε με θέματα που δεν μπαίνουν στις δημοσιονομικές προοπτικές. Ε, Μιλήσαμε για πολλά θέματα, για τις την οικονομική κρίση και για χίλια άλλα ακόμα, αλλά δυστυχώς ε, στην τελική έκθεση δεν αποκρισταλώνονται αυτά. Αλλά νομίζω ότι τα περισσότερα αιτήματα, οι διεκδικήσεις της Επιτροπής σας ελήφθηκαν υπόψη. Θα δούμε στη συνέχεια τη συζήτηση αν σφάλω με διορθώστε. Για να μπω τώρα λίγο στην ουσία, μια μικρή σύνοψη των όσων συμπεριλάβαμε στην έκθεσή μας. Ένα από τα βασικά που λέμε ε, ως προς την ανάπτυξη και την ανάπτυξη ψυχιακή βοήθεια και το κεφάλαιο 4 τη συνολικής Ευρώπης είναι ότι υποχρηματοδοτείται αυτή η κατάσταση και μάλιστα η κατάσταση είναι χρόνια στο έλλειμμα παντού στον κοινοτικό προπολογισμό, αλλά ιδιαίτερα στο τίτλο 4 που έχει σχέση με την Ευρώπη και την παρουσία της στον κόσμο. Ε, το έλλειμμα αυτό είναι και χρόνιο όσο και ανησυχητικό. Επίσης ε, λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μεγάλο πρόβλημα ευελιξίας ε, στον προπολογισμό και αυτό το λέμε και κυρίως προς το Συμβούλιο, όχι επειδή δεν έχουμε μέσα ευελιξίας, αλλά επειδή ποτέ δεν θέλει να τα κινητοποιεί το Συμβούλιο. Και αυτό είναι σοβαρό, ιδιαίτερα όταν δούμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε εσείς στην Επιτροπή σας και διαπραγματεύεστε, γιατί είναι έκτακτα όλα, απρόβλεπτα. Ε, καταστροφές, θεομηνίες, κρίσεις ε, σε αναδυόμενες χώρες, ανάγκες που δεν μπορεί κανείς να προβλέψει για την επόμενη δεκαετία. Γι' αυτό ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το Συμβούλιο να τα λαμβάνουν υπόψη και να χρησιμοποιούν αυτά τα μέσα ευελιξίας, τα οποία διαθέτουμε μεν, πριν όμως ποτέ δεν χρησιμοποιούμε. Και επίσης δεν λέμε μόνο περισσότερα χρήματα, αλλά περισσότερο περιθώριο. Δηλαδή ακόμα και χρήματα που ε, δεν θα έχουν εγγραφεί στον προπολογισμό να είναι στη διάθεσή μας για να το εκταμιεύσουμε. Αυτό γενικά, ε, ως προς τα αιτήματα πάντα. Για την καταπολέμηση της ένδυας, λέμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το 2015 είναι πολύ κοντά μας και οι αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας δεν πρόκειται να επιτευχθούν εκτός ε, εάν βάλουμε ε, το χέρι στην τσέπη και βγάλουμε τα χρήματα που χρειαζόμαστε. Επίσης, ε, λέμε ότι συνεχίζουμε να έχουμε ως στόχο το 0,7% ως επίσημη κρατική αναπτυξιακή βοήθεια και θέλουμε περισσότερα να κάνουμε. Γιατί αυτού του στόχου του έχει θέσει όχι μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και τα 27 κράτη-μέλη και το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τι δεσμεύσει που απορρέουν από την Κοπεχάγη και την Κανκούν για το περιβάλλον. Επίση, ζητούμε στον κοινοτικό προϋπολογισμό να εγγραφεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο ανάπτυξη, να ενταχθεί στον προπολογισμό. Αυτό είναι πάγιο αίτημα, θα θυμάστε, και ιστορικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη Επιτροπή σα. Σε ό,τι αφορά τις αναδυόμενες χώρες, ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εντάσει εναλλακτικά συστήματα για την αναπτυξιακή συνεργασία με τις χώρες αυτές και να μπορούν να προσαρμόζουν τις πολιτικές τους. Και επίσης να μελετήσει τη δυνατότητα κινητοποίησης ενός νέου μέσου ε, για δραστηριότητες που δεν είναι επίσημα χρηματοδοτούμενες από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, αλλά μπορούν να συνδυάσουν, να συγκεράσουν τα αμοιβέ συμφέροντα των χωρών μας. Παράδειγμα, ε, ανθρωπιστική βοήθεια. Βεβαίως υποστηρίζουμε και προφανώς και τονίζουμε και πάλι τη σημασία που έχει η ανθρωπιστική βοήθεια και για άλλη μια φορά ζητούμε χρηματοδότηση. Ουσιαστικά τι κάνει η έκθεση. Τονίζει πόσο σημαντικέ είναι οι πολιτικές που χαράσουμε και ακολουθούμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πάντα λέμε ότι τα χρήματα δεν φτάνουν. Άρα χρειάζεται μεγαλύτερη πρικοδότηση. Και τελειώνω με τα χρηματοδοτικά μέσα και τα καινοτόμα μέσα. Θα χρειάστηκε να είμαστε πολύ πιο συγκεκριμένοι, πολύ περισσότερο από ό,τι θα θέλαμε. Ξέρω ότι η γνωμοδότησή σας της Επιτροπής Ανάπτυξης έμπαινε σε χωράφια που δεν ήταν δική μας ε, αρμοδιότητα Πάντως κάναμε αναφορά εκεί και στους ιδίους πόρους και στο φόρο χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Δεν λέμε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να αφιερωθούν αυτά τα έσοδα στην αναπτυξιακή βοήθεια ή στους στόχους της χιλιετίας, αλλά είναι προφανές αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση καταφέρει να αυξήσει τους πόρους και έχει περισσότερα έσοδα, προφανέστατα θα ε, μπορεί να χρηματοδοτεί και την αναπτυξιακή πολιτική πολύ καλύτερα ή άλλη πολιτική γιατί θα είχαμε χρήματα που θα περίσσευαν για την αναπτυξιακή πολιτική. Τελικά ο στόχος είναι να αυξηθεί ε, η κατηγορία των εσόδων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορεί να δαπανά και περισσότερο και καλύτερα και για την αναπτυξιακή βοήθεια. Αυτά δεν θα επεκταθώ περισσότερο. Δεν ξέρω αν έχετε ερωτήσεις σε ιδιαίτερα ή αν έρθει ο εισηγητής, γιατί εγώ είμαι μια απλή σκιώδης εισηγήτρια. Αυτά. Ευχαριστώ. Je passe la parole à Monsieur Θα δώσω το λόγο στον κύριο Γκέρενς. Ευχαριστώ πολύ. Θα κρατήσω την τελευταία φράση. Ε, κοιτάξτε, εγώ τελικά είμαι απλώς ο αντικαταστάτης του κυρίου Τις Μπέρμαν ο οποίος ήδη στο εμπαρόδο είναι και αντικατάστατος. Εν πάση περιπτώσει, ελπίζω ότι θα του μεταφερθούν τα πράγματα ακριβώς όπως τα είπα, γιατί δεν θέλω να μπερδευτούν η σχέση μου με τον ε, Τάις Μπέρμαν. Ο τρόπος με τον οποίο φέρθηκε η Επιτροπή Σούρε στην ε, Επιτροπή ανάπτυξης ε, δεν ήταν και ο χειρότερος δυνατός. Ε, ελήφθησαν υπόψη ε, κάποιες ιδέες μας, άλλες και προτάσεις μας, άλλες όχι. Πρέπει να πω πάντως ότι οι γνωμοδοτήσεις των διαφόρων επιτροπών δεν ελήφθησαν όλες υπόψη. Δηλαδή δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι εμείς υπέστημε διακριτική μεταχείριση ή ότι ε, μόνο εναντίον μας ας πούμε ε, ελήφθησαν έτσι αυτές οι θέσεις. Λοιπόν, στο κείμενο αναφέρονται κάποιες ε, ιδέες τις οποίες η Επιτροπή μας είχε κοινοποιήσει στην ΣΟΥΡΕ κάποιες δεσμεύσεις σχετικά με τους στόχους της χιλιετίας. Επίσης η αποτελεσματικότητα της βοήθειας που αναφέρεται στη δήλωση των Παρισίων. Ένα σημείο το οποίο μας είναι προσφυλές και το οποίο καταδείξαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είμαστε οι πρώτοι που το κάναμε, είναι η αρχή της προσθετικότητας των των ε, πόρων που θα δοθούν για την ε, μετρίαση το, της ε, κλιματικής αλλαγής στις αναπτυσσόμενες χώρες. Είπαμε ότι οι διάφοροι πόροι θα πρέπει να δοθούν σε ένα... θα πρέπει να δίδονται με προσθετικό τρόπο. Και ότι θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια να ληφθούν υπόψη και οι αναδυόμενες και οι νεοαναδυθήσεις οικονομίες, καθώς επίσης και δυνατότητα μεταφοράς ε, ε, κεφαλαίων που δεν θα έχουν δαπανηθεί. Πάντως διαπιστώνω ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν μας άκουσε η Επιτροπή Σούρε και ότι δεν έλαβαν υπόψη τις προτάσεις μας. Euh, Ένα σημείο το οποίο αφορά μάλιστα και εντάσσεται σε μια συζήτηση που κάναμε στην αρχή της ε, συνεδρίας μας και που αφορά στην ανθρωπιστική βοήθεια διαπιστώνουμε ότι αντιμετωπίζουμε όλο και περισσότερες φυσικές καταστροφές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξοδεύει πολλά έτσι ώστε να βοηθήσει σε αυτές τις περιπτώσεις. Και εμείς επιμείναμε στην ουδετερότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Ουδετερότητα δεν είναι ο πλέον προσήκον όρος, αμεροληψία θα έλεγα εγώ καλύτερα. Δεν μπορεί κανείς, ε, δηλαδή μπορούμε να μην είμαστε ουδέτεροι απέναντι σε αιμοσταγείς ε, δικτάτορες, ε, μπορούμε να είμαστε αμερόληπτοι, όπως ο Καντάφη, μπορούμε να είμαστε αμερόληπτοι όμως. Δηλαδή μπορούμε να προχωρήσουμε σε ανθρωπιστική βοήθεια προς τη χώρα του χωρίς αυτό να αλλάζει την άποψη που έχω για τον άνθρωπο αυτό και την οποία μόλις εξέφρασα. Και πρόκειται και για μια έτσι γενική σκέψη, ε, γιατί πρέπει να σας πω ότι εμείς ε, είπαμε ότι τα προβλήματα θα πρέπει να, να αντιμετωπιστούν ε, σφαιρικά και συνεκτικά. Και επομένως αυτές ήταν οι ιδέες οι οποίες θεωρώ ότι θα έπρεπε να θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη αυτό το 0,7 ε, η τυπλοποίηση του Ταμείου ε, Α, και να πω επίσης ε, ότι και ο πρόεδρος Λαμασούρ de, de... ανέφερε ότι ε, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ε, να κάνουν ε, κάποια κράτη πολιτική πέραν του προϋπολογισμού. Δηλαδή, κυρίως αναφέρθηκε στο Ταμείο που ε, προσπαθεί να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες κυρίως χώρες ε, να καταπολεμήσουν ε, τις καταστροφικές συνέπειες των, της κλιματικής αλλαγής. και ότι η, το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης με αυτό το σκεπτικό ε, θα αποκτούσε μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. Αυτά. Δεν υπάρχει και τίποτα ιδιαίτερα νέο σε αυτά που μόλις σας είπα. Δεν μπορώ να πω αν οι ιδέε ε, ε, θα έλεγα ότι ήταν κοινότοπες. Δεν θέλω όμως όλε αυτή την επίκριση. Τέλος, ένας συνάδελφος μου είπε ότι η πρωτότυπε. εγω μαλλον θα ελεγα οτι ηταν κοινοτοπε δεν θελω ομως να ξεκινησει ετσι μια ολοκληρη ιδέα είναι μια κοινότοπη ιδέα που είμαστε οι πρώτοι που την εκφράσαμε. Επομένως δεν μας ενδιαφέρει αν είναι τα πρωτότυπη ή όχι η ιδέα. Μας ενδιαφέρει να την ε, εφαρμόσουμε σωστά με την ελπίδα ότι στο τέλος ε, της συζήτησης κάποιος ηθήνων θα μας ακούσει. Ε, και σίγουρα όσον αφορά την εγγραφή στο προπολογισμό, σίγουρα δεν θα το κάνει το Συμβούλιο στη θέση μας. Επομένως εδώ να ευχαριστήσω και την εκπρόσωπο της ΣΟΥΡΕ και νομίζω ότι δεν έχουμε μεγάλες ε, διαφορές. Ε, είμαστε σε ίδιο μήκος κύματος. Νομίζω ότι πρέπει να χαρούμε γιατί η συνεργασία όσον αφορά τα θέματα ανάπτυξης και στην Επιτροπή ΣΟΥΡ και στην Επιτροπή προπολογισμών είναι σημαντική. Και ξέρετε δεν είναι απολύτως προφανής. Γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι για αυτή την ε, ταυτοσημεία απόψεων ε, σε ένα τόσο διαφορετικό περιβάλλον. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε λίγα λεπτά στη διάθεσή μας. Στην κυρία Κέλλερ θα δώσω το λόγο και μετά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ. You have a bit of a more critical, um ευχαριστώ. Εγώ είμαι λίγο πιο ε, επικριτική, ίσως είμαι και υπερβολικά φιλόδοξη. Βρίσκω ότι είναι λυπηρό το γεγονός ότι καμιά από τις τροπολογίες μας δεν έγινε δεκτή. Τώρα θα έχουμε λοιπόν ένα κεφάλαιο στην έκθεση Σούρε για θέματα ανάπτυξης και ναι βέβαια λέτε περίπου τα ίδια πράγματα με αυτά που λέμε εμείς, αλλά είναι πολύ γενικό. Εάν δεν χρειάζεται τη γνωμοδότηση της ειδική Επιτροπής, αν βάλετε μόνο τα πράγματα τα οποία ε, έχετε ε, καταλήξει εσείς, νομίζω ότι αυτό είναι κρίμα. Το ίδιο θα συμβεί και με άλλες ε, κοινοβουλευτικές επιτροπές, που επίσης και εκεί οι απόψεις τους δεν αναγνωρίστηκαν. Και έχουμε γενικά το πρόβλημα της γνωμοδοτήσης διότι για μας την Επιτροπή Ανάπτυξης οι γνωμοδοτήσει είναι το πιο σημαντικό εργαλείο για να προωθήσουμε τις ε, πολιτικές μας. Κάνουμε γνωμοδοτήσεις για την Επιτροπή Αλίας, για την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου κλπ. Και το βλέπουμε ξανά και ξανά ότι αγνοούνται πλήρως οι θέσεις μας. Μπορούμε να καταθέτουμε τροπολογίες, εμείς οι ίδιοι δηλαδή ατομικά, αλλά η ιδέα γενικά της γνωμοδότησης είναι ότι την στηρίζει ολόκληρη η Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Αλλά οι αρμόδιες επί της συχνά της αγνών. Και αυτό είναι πρόβλημα, διότι δεν μπορούμε με τον τρόπο αυτό ούτε να υλοποιήσουμε την φιλοδοξία μας, να έχουμε δηλαδή να είμαστε συνεκτικοί στην προσέγγιση μας για την πολιτική ανάπτυξη. Δεν ξέρω βέβαια τι μπορεί να γίνει προκειμένου, γιατί η συζήτηση αυτή πρέπει να γίνει και γενικότερα. Αν όμως δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς αποτελεσματικά τον μηχανισμό των γνωμοτήσεων, τότε τι να κάνουμε. Μήπως να κάνουμε μια απεργία, να σταματήσουμε να γράφουμε γνωμοδοτήσεις, για να δείξουμε ότι εν πάση περιπτώσει μας απασχολούν στα σοβαρά. Δεν ξέρω αν είναι πραγματικά κατάλληλος ο τρόπος αυτός. Κάνω τέλος πάντων, ίσως να κάνω την πρόταση αυτή. Το, για το θέμα τώρα του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Αυτό έχουμε τώρα και με αυτό θα αναγκαστούμε να εργαστούμε. Θα παρακολουθούμε προσεκτικά τις λεπτομερείς προτάσεις οι οποίες θα προκύψουν από την εργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα τις εξετάσουμε λοιπόν προσεκτικά και όχι μόνο για την κατηγορία 4, όπου θα μπει η αναπτυξιακή βοήθεια, αλλά και τους άλλους τομείς όπου συχνά έχουν σχέση με ε, την ανάπτυξη. Για παράδειγμα, προϋπολογισμός της ε, ε, Επιτροπής Γεωργίας ή της Επιτροπής Θεμελιωδών Ελευθεριών. Δεν θα σταματήσουμε λοιπόν να κοιτάζουμε και πέραν των ορίων αρμοδιότητας της δικής μας Επιτροπής για να παρακολουθούμε το ότι εξελίσσεται. Μάλιστα, πριν δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πω ότι, λαμβάνοντας το λόγο εγώ, η ιδία ότι είναι γεγονός ότι η κατάληξη είναι καλή, αλλά πάντω οι θέσει μας δεν λήφθηκαν υπόψη. Θα συμφωνήσω με την κυρία Κέλλερ, διότι αυτό είναι λυπηρό, διότι φαίνεται σαν να μην εξυπηρετεί απολύτως τίποτα η προσπάθεια μας αυτή. Εγώ θεωρώ λοιπόν επίσης ότι πρέπει να σκεφτούμε λίγο τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε η εργασία μας και να ακούγεται και να περιλαμβάνεται διότι δεν είναι και νορμάλ αυτό. Επειδή έχει γίνει πάντα μέχρι τώρα έτσι δεν σημαίνει ότι έτσι πρέπει να συνεχιστεί. Τώρα λοιπόν σα τα είπα, θα δώσω το λόγο στον κύριο Άτλαν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συντονίζεται απολύτω ε, με τις προτάσεις τη έκθεση, η οποία μπορεί να μην είναι καινοτόμα από το α μέχρι το ω, αλλά είναι ποτισμένη από ε, ορθολογισμό ε, και ακριβώς αναφέρει όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να αποτελέσουν βάση της ε, αναθεώρησης ε, των υπαρχόντων μηχανισμών και εργαλείων. Αναφέρθηκαν ήδη κάποιοι βουλευτές σε μια σειρά θεμάτων που μας φέρονται σημαντικά. Πρώτον, θα πρέπει να παραμείνει ενιαίο το κεφάλαιο 4, έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που έχουν βάσει της συνθήκη της Λισαβόνας. Δεύτερη αρχή η αρχή της προσθετικότητας των πόρων. Συμμεριζόμαστε απολύτως την άποψη αυτή. Ε, πραγματικά θα πρέπει να υπάρξει στενός συσχετισμός ανάμεσα σε κάθε νέα ε, προτεραιότητα και τον αντίστοιχο ε, πόρο. Και αυτό έτσι ώστε να μην ε, δυναμητιστούν οι ήδη, πολιετή, οι ήδη υπάρχοντες σχεδιασμοί. Επίσης, βάσει των περισσότερων εργαλείων. Ε, εκεί συμμεριζόμαστε απολύτω τον στόχο του 0,7 και θα πρέπει να διατηρηθεί ο στόχο αυτό, και να είμαστε πολύ ρεαλιστές ε, όσον αφορά τον ορίζοντα 2011. Επίσης, η αρχή της αποτελεσματικότητας ε, της ε, βοήθειας. Ε, επίσης, η επικύρωση των στόχων της δήλωσης των Παρισίων. Πρέπει να πούμε ότι αυτή είναι μια καλή βάση, έστω και αν μέχρι τώρα δεν έχουμε επιτύχει σε όλα, πάντως πιστεύω ότι θα αποτελέσει μια καλή βάση για τον ορισμό των εργαλείων. Επίσης, όσον αφορά την ε, αποτελεσματικότητα της βοήθειας θα πρέπει να δούμε το υποσημείο καλή συνεργασία με τα κράτη-μέλη που θα αποτελέσει φυσικά αντικείμενο συγκεκριμένων προτάσεων της Κομισιόν. Συμμεριζόμαστε επίσης πλήρως την άποψη που εκφράζει η έκθεση όσον αφορά την ιδιαιτερότητα της ε, Ένωσης, όσον αφορά την γειτονία και κυρίως ε, όσον αφορά την στρατηγική προτεραιότητα η οποία θα πρέπει να δοθεί στην καλή διακυβέρνηση, στην ανθρώπινα δικαιώματα ε, και την προστασία των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτή η ιδέα των, της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει οπωσδήποτε να ενισχυθεί. Όσον αφορά τώρα την ε, προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία. Πρόκειται για μια αξία η οποία έχει ήδη καταδειχθεί και όσον αφορά ε, τη διεύρυνση και όσον αφορά την ε, γειτονία. Πιστεύουμε ότι η κοινοτική δράση δεν θα πρέπει να είναι μονάχα ποσοτική, αλλά θα πρέπει να είναι και πολιτική. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ε, λαμβάνοντας υπόψη κυρίως όσον αφορά την ελευθερία κυκλοφορίας αγαθών, ε, αγαθών κεφαλαίων, ε, προσώπων, ε, δημοκρατία, εκδημοκρατισμό κτλ. Ε, μιλάμε κυρίως για ποιοτικέ πολιτικές και όχι ποσοτικές. Επίσης, η Κομισιόν στηρίζει πλήρως τη θέση της έκθεσης σχετικά με την ανάγκη αύξησης της ευελιξίας του προϋπολογισμού ευελιξία μεταξύ των κεφαλαίων έτσι ώστε οι υπεύθυνοι της, Υπηρεσία της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης να μην είναι οι μόνοι που θα πρέπει να επομιστούν το βάρος των ε, κρίσεων και των έκτακτων καταστάσεων. Ας πούμε, η μετανάστευση αφορά και τις εσωτερικές πολιτικές κοινότητας. Είπαμε λοιπόν ευελιξία και στο κεφάλαιο 4, αλλά ε, με κάποια όρια έτσι ώστε να μην τεθεί ένα αμφιβόλο η αρχή της, ε, ε, του πολιετού προγραμματισμού αναφορά αφορά την διεύρυνση και την γειτονία. Τέλος, ευελιξία στα ίδια τα εργαλεία. Ας πούμε, το εργαλείο ΕΙΠΑ για το οποίο έχει προγραμματιστεί συγκεκριμένο κονδύλι. Ε, αυτό μπορεί να ισχύει αντίστροφα και με ολίσθηση ε, των πόρων που θα δοθούν σε μια χώρα σε περίπτωση που δεν θα έχει η χώρα αυτή ε, τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ε, σε 30 δεύτερα που μου μένουν θα ήθελα να ε, πω ότι όσον αφορά την εταιρική σχέση για ενισχυμένη βοήθεια προς τις αναπτυσσόμενες χώρες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει ευρύτερη βάση από ότι ε, το παρόν εργαλείο του ICI. Θα υπάρξει επομένως αναθεώρηση του παρόντος εργαλείου. Πολύ σύντομα, πολύ σύντομα κι εγώ. Εγώ δεν θέλω να είμαι τόσο αρνητικό όσο η συνάδελφο Κέλλερ. Νομίζω ότι πολλά στοιχεία πήρε από εμά η, Ευρωπαϊκή, η Επιτροπή Σούρε. Εγώ πιστεύω ότι η Επιτροπή συνεννοήθηκε μαζί μας πριν από την σύνταξη της θελητής έκθεσης και νομίζω ότι τα δύο τελευταία χρόνια ασχοληθήκαμε με θέματα τα οποία τελικά ενέταξε η Σούρα στην έκθεσή της. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να είμαστε τόσο υπερβολικοί σε αυτά τα σημεία, δηλαδή να μην κάνουμε και απεργία για αυτό το θέμα. Εγώ θα έκανα απεργία για κάποια άλλα θέματα. Εντάξει, αυτή είναι και η δική μου άποψη. Ναι, και βλέποντας λίγο για την κατάσταση, ε, εδώ <laughs> νομίζω ότι δεν είναι και πολύ τιμητική η κατάσταση. Ε, δηλαδή ζητάμε δεξιά και αριστερά φωνασκούμε λέγοντας θέλουμε περισσότερα, ε, περισσότερα δικαιώματα και τελικά είμαστε τρεις και ο κούκος. Και πραγματικά εάν άφηνε τον εαυτό μου να μιλήσει όπως θα ήθελε, ε, δεν θα μπορούσαν να δημοσιευθούν τα λόγια μου. Θέλετε να τελειώσετε, να ολοκληρώσετε τη συζήτηση. Ναι, ναι, ένα λεπτάκι μόνο. Ε, Έλεγε ο προλαλής σας και έχει δίκιο ότι στην έκθεσή μας πράγματι συμπεριλάβαμε τις μεγάλες προτεραιότητες και τις στρατηγικές γραμμές και τα μεγάλα αιτήματα της δικής σας Επιτροπής. Είναι γεγονός ότι δεν επισυνάφθηκαν ε, οι γνωμοδοτήσεις στην έκθεση, δεν ε, θεωρήθηκαν παράρτημα, αλλά έχουν ενταχθεί στην έκθεση οι υπόλοιπε γνωμοδοτήσει των υπόλοιπων επιτροπών. Κάποιος είπε η κυρία Κέλλερ προηγουμένως ότι δεν λάβαμε υπόψη μας τροπολογίες. Μα ήταν 1041 οι τροπολογίες. Όλες τις μελετήσαμε, ε, τις εξετάσαμε και ομαδοποιήσαμε τις περισσότερες σε συμβιβαστικές. Και τις υπόλοιπες τις ψηφίσαμε. Τώρα το θέμα είναι ότι ορισμένες επιτροπές ή ορισμένοι βουλευτές έκαναν τροπολογίες που δεν υπερψήφισε η πλειοψηφία των βουλευτών. Αυτό συνέβη και στην ομάδα μου και σε μένα προσωπικά. Κατέθεσα τροπολογίες που δεν εγκρίθηκαν. Ε, τι να κάνουμε, έτσι έχει το παιχνίδι των κοινοβουλευτικών επιτροπών και της Ολομέλειας. Άλλες ε, τροπολογίες κερδίζουμε, άλλες χάνουμε. Τι να κάνουμε. Και εγώ είχα μεγάλη φιλοδοξία από την έκθεση, αλλά εκτός από τη συνένεση όλων των πολιτικών ομάδων, ε, ζητούσε ε, και ενίσχυση και υποστηρίχθηκε από το ΕΛΚ, τους σοσιαλιστές, τους φιλελεύθερους και τους πρασίνους. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Διακόπτεται η συνεδρίαση, θα συνεχιστεί αύριο στις 10, ενώ στις 9 θα συνεδριάσουν οι συντονιστές στην παρούσα ε, αίθουσα. Καλό σας βράδυ και σας ευχαριστώ.